Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Καλώς ήρθατε μετά από ε, τις καλοκαιρινές διακοπές. Μπορούμε να περάσουμε στην υιοθέτηση της ημερήσιας διάταξης. Ωραία. Τώρα όσον αφορά τις ανακοινώσεις, ως συνήθως θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η συνάντηση ε, μεταδίδεται online και τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στη σελίδα της ΣΥΜΚΟ. Όσον αφορά τα πρακτικά της 13ης και 14ης Ιουλίου θα παρουσιαστούν την 26η Σεπτεμβρίου, οπότε δεν χρειάζεται να τα ε, υιοθετήσουμε σήμερα. Και δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση σχετικά με τους τριμερείς διαλόγους και τις εκδηλώσεις. Ελπίζω όλοι να είχαν ένα καλό καλοκαιρινό διάλειμμα. Τώρα όσον αφορά την ε, έγκριση ε, για τα μηχανοκίνητα οχήματα. Αυτό αναβάλλεται, οπότε περνάμε κατευθείαν στην παρουσίαση από την πλευρά της ε, Κομισιόν σχετικά με την πρόταση που αφορά τα συμβόλαια για τις ε, ηλεκτρονικές πωλήσει, ε, το οποίο αφορά συγκεκριμένα τα πρώτα αποτελέσματα του ε, Refit. Η συγκεκριτής είναι ο Πασκάλ Αχιμού. Ευχαριστώ Πασκάλ. Και θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι λάβαμε επιστολή από την πλευρά της Κομισιόν τον Αύγουστο που ε, περιέχει ορισμένα στοιχεία για, με τα δεδομένα για την αγορά αγωθών, ε, τα οποία έχουν αγοραστεί πρόσωπο κατά πρόσωπο, αλλά και εξ αποστάσεως, καθώς επίσης ε, και άλλα υποστηρικτικά δεδομένα, τα οποία διατίθενται στην ιστοσελίδα μας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Βερόνικα Μαφρέντι από τον ε, τομέα και των ελωτών ε, της ε, Κομισιόν που θα παρουσιάσει τα πρώτα αποτελέσματα. Βερόνικα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους μια καλή αρχή. Ξεκινάει ουσιαστικά η καινούρια περίοδος για όλους. Η σημερινή παρουσίαση ελπίζω να είναι ένα ενδιαφέρον ορεκτικό, γιατί μας περιμένει πολύ μπροστά, πολλή δουλειά μπροστά μας, για να μπορέσουμε να πετύχουμε να υπάρχουν σωστά, κατάλληλα, λειτουργικά μέσα ε, υπεράσπιση των καρναλωτών ε, σε ό,τι αφορά την πώληση αγαθών επιγραμμικά αλλά και μη επιγραμμικά. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ στους πολιτικούς στόχους, καταρχήν, πίσω από την πρόταση την οποία εγκρίναμε στις 9 Δεκεμβρίου του 2015. Εγκρίναμε ένα πακέτο προτάσεων, μια πρόταση οδηγίας που θα δίνει στους καταναλωτές ε, αποτελεσματικά ε, ένδικα μέσα ε, όταν έχουμε ελαττωματικά προϊόντα και υπηρεσίες και επίσης ε, μια οδηγία για ε, τα ε, απτά αγαθά σε ψηφιακή όμως πώληση. Γιατί δίνουμε έμφαση στο ψηφιακό σκέλος. Έχουν γίνει σημαντικές εργασίες για την προετοιμασία της στρατηγικής για την ψηφιακή αγορά και κατά την προπαρασκευή αυτή έγινε σαφές ότι υπάρχουν μεγάλες ε, δυνατότητες βελτίωσης, μεγάλες δυνατότητες επέκτασης και ανάπτυξης. Επίσης, κατέστησα σαφές από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι επιχειρήσεις, οι καταναλωτές, ε, οι εθνικές αρχές, ε, κατέστησε σαφές λοιπόν ότι υπάρχει μια έκκληση ή δυνατόν να έχουμε τα ίδια μέσα αντίδρασης για τους καταναλωτές και επιγραμμικά και μη επιγραμμικά και συμβατικά. Έγινε λοιπόν μια προσπάθεια να τροφοδοτήσουμε την νομοθετική διαδικασία που θα ξεκινούσε με περαιτέρω στοιχεία για το πώς η παρούσα οδηγία για τις εγγύησεις στους καταναλωτές εφαρμόζεται ε, και μπορεί να εφαρμοστεί και επιγραμμικά έτσι ώστε να υπάρξει μια ευθυγράμμιση δηλαδή των κανόνων σε ό,τι αφορά τα μέσα αντίδρασης. Τα μέσα προστασία του καταναλωτή. Και τώρα είναι η στιγμή της αλήθειας για κάποιο τρόπο. Ερχόμαστε με πάσα ειλικρίνεια να σας παρουσιάσουμε τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μα. Θέλω να υπογραμμίσω όμως, όπως είπε και η Επίτροπο στην επιστολή που έστειλε αρχές Αυγούστου, Βεβαίω φαντάζομαι ότι αυτή την επιστολή τη λάβατε κάπου σε κάποια παραλία, ε, να πούμε πάντως ότι τα δεδομένα αυτά ακόμα τα επεξεργαζόμαστε, τα εξετάζουμε και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρετε ότι το REFIT, το REFIT ε, είναι μια διαδικασία που αποτελεί μέρος των καθητήριων γραμμών για την καλύτερη νομοθεσία. Χρειάζεται λοιπόν η κατάλληλη διαφούλευση όλων των ε, εμπλεκομένων πλευρών και εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα. Σκεφτήκαμε πάντως ότι καλό θα ήταν να σας παρουσιάσουμε ε, ποιες είναι οι γενικές τάσεις διότι αυτές είναι που θα επιβεβαιωθούν και από την τελική έκθεση την οποία θα μοιραστούμε μαζί σας τον Σεπτέμβριο. Περνάμε λοιπόν τώρα στην επόμενη διαφάνεια. Γνωρίζετε ότι το REFIT είναι μια, ένα ευρύτερο εγχείρημα. Η οδηγία για τις εγγύες των καταναλωτών είναι μία από τις έξι οδηγίες που εξετάζονται αυτή τη στιγμή. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο εξετάζει ε, σημαντικές και εναρμονισμένες νομοθεσίες ε, για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές παραδείγματος χάρη, η σχετική οδηγία. Ε, δεν υπάρχει όμως επαρκής εναρμόνιση ε, σε κάποιες άλλες οδηγίες για τις προσφυγές, για τις διαταγές πληρωμής. Με βάση τη δέσμευση που αναλάβαμε το δεκαετία του 2015 έχουμε βάλει πρώτα χρονικά τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την οδηγία για την προστασία των καταναλωτών. Και βεβαίως ε, θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας έτσι ώστε να σας δίνουμε συνεχώς τα πιο ε, επίκαιρα στοιχεία, τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το θέμα αυτό. Πάμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια για να σας δείξουμε λίγο τι έχουμε κάνει σε επίπεδο έρευνα έως τώρα. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτά τα πρώτα δεδομένα έχουν ένα σημαντικό στοιχείο. Ε, προέρχονται δηλαδή απευθείας ε, από τους ενδιαφερόμενους. Ε, σε επίπεδο καταναλωτών μιλήσαμε με 23.500 καταναλωτές στα 28 κράτη-μέλη συν την Ορβηγία και την Ισλανδία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε ένα σημαντικό αριθμό πραγματικών παραδειγμάτων που μας την άποψή τους. Σε επίπεδο τώρα γενοπολιτών έχουμε ένα πολύ πιο μικρό αριθμό, 375 όντως, σε 15 κρατη όμως μόνο. Μιλάμε για 185 πραγματικές, πραγματικά μικρές επιχειρήσεις, κάτω από 10 ε, ε, εργαζόμενοι. 153 μικρές επιχειρήσεις και 37 μεσαίες. είναι δύσκολο ε, να φτάσει η Κομισιόν σε επαφή με, την, ε, ε, με τους απλούς πολίτες και αυτούς που πραγματικά επιτόπου επηρεάζονται τις πολιτικές αυτές. Πάντως συνεχίζουμε εμείς σε επίπεδο ΙΜΚΟ να προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτά τα στοιχεία. Προσπαθούμε να ανοίξουμε διάβλους επικοινωνίας και με τι επιχειρήσεις. Περνάμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια για να, για να εξηγήσουμε καταρχήν την οικονομική σημασία της ευθυγράμμισης των κανόνων ε, για τις επιγραμμικές πωλήσεις και τις μη επιγραμμικές πωλήσει. Να δώσουμε κάποια στοιχεία πρώτα. Πρώτα απ' όλα, θα γνωρίζετε ίσως ότι στην ευρωπαϊκή οικονομία έχουμε περίπου ...1,2 εκατομμύρια δινοπολιτές το 35% δηλαδή του συνόλου λιανοπολιτών πολλούν και εξ και ε, συμβατικά. Είναι ένα σημαντικό λοιπόν ποσοστό της οικονομίας μας, πολλοί επιχειρηματίες, πολλοί έμποροι θα επηρεαστούν άμεσα από τις επιλογές των νομοθετών για το κατά πόσο τελικά θα είναι ήδη ρυθμιστικό πλαίσιο και για τις επιγραμμικές πωλήσει και για τις μη επιγραμμικές πωλήσει. από αυτούς που πολλούν συμβατικά 42% είναι 56% του συνόλου αυτοί που πολλούν συμβατικά, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας, από αυτούς λοιπόν το 56%, το 42% λέει ότι το γεγονός ότι υπάρχουν ε, αποκλίνοντες κανόνες ε, αποτελεί σημαντικό ή αρκετά σημαντικό εμπόδιο στη φιλοδοξία τους να αναπτυχθούν περαιτέρω διασυνοριακά. Ε, στην αξιολόγηση αντικτύπου στην αντιπρόταση για τα ψηφιακά είχαμε πει ότι ο αριθμός αυτός είναι 46% σε ό,τι αφορά τους λιανοπολιτές επιγραμμικά δεν είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Βλέπετε ότι είναι ένα μεγάλο αριθμό των πολιτών, είτε πολλούν συμβατικά είτε επιγραμμικά, ε, που έχουν εντοπίσει αυτό το πρόβλημα. Πάμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια για να δούμε τι γίνεται τώρα από πλευρά καταναλωτών. Εδώ διαπιστώνουμε ότι οι καταναλωτέ, αυτοί οι περίφημοι 23.500 καταναλωτέ, μα λένε ότι πάνω μάλλον πάνω από, πάνω από το 3% συνήθως αγοράζουν συμβατικά τα προϊόντα στο μαγαζί. Είναι μόλις 49% σε ό,τι αφορά τις επιγραμμικές πωλήσει και σε ό,τι αφορά το διασυνοριακό εμπόριο ξαφνικά το ποσοστό πέφτει πολύ, μόλις 11%. Και μόλις 17% αγοράζουν επιγραμμικά από μια άλλη χώρα της Ένωσης. Ακόμα δηλαδή και όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό, ε, οι άνθρωποι αυτοί ε, δεν ψωνίζουν πολύ. Βεβαίως όλοι είχαμε κάποια ευχάριστη εμπειρία αυτό το καλοκαίρι, αλλά υπάρχει έτσι μια κάποια έλλειψη εμπιστοσύνη όταν κάποιος πάει να αγοράσει ένα προϊόν σε μια άλλη χώρα. Και βεβαίως έχουμε το θέμα των ε, βιώσιμων αγαθών, έτσι μόλις 5% καταναλωτών έχουν συγγνώμη, 5% καταναλωτών έχουν ταξιδέψει ε, συχνά ή αρκετά συχνά σε μια άλλη χώρα της Ένωσης για να αγοράσουν αυτά τα προϊόντα και 30% το έχουν κάνει κάποιες φορές ή σπάνια. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά. Το οποίο βέβαια προφανώς ε, έχει εξηγήσει. Δεν θα πήγαινα ούτε εγώ σε μια άλλη χώρα να αγοράσω ένα ψυγείο. Όμως ε, όταν μιλάμε για κάποιο iPhone ή για κάποιο άλλο ε, κάποια άλλη συσκευή IT γιατί κάποιος να μην προσπαθήσει να μεταλλευτεί κάποια πιο φθηνή τιμή ή κάποια μεγαλύτερη γκάμα ε, επιλογών σε μια άλλη χώρα. Εδώ πάλι ενδεχομένως να υπάρχει μια ανασφάλεια σε ό,τι αφορά το ποιο καθεστώς ε, ισχύει, ποιο είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο όταν κάτι δεν πάει καλά. Εάν δείτε τα παρατήματα που σας στείλαμε, θα διαπιστώσετε ότι πολλοί καταναλωτές λένε ότι το γεγονός ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν ένα διαφορετικό ρυθμιστικό πλαίσιο ε, παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην απόφαση που παίρνουν. Είναι από του πιο σημαντικούς παράγοντες να λάβουν την απόφασή τους. Πάμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπετε Ποιε είναι οι βασικές ε, πολιτικές επιλογές ε, τις οποίε έχουν μπροστά μα ως Κοινοβούλιο και ω Συμβούλιο βέβαια. Πρώτα απ' όλα εξετάζουμε πώς συμπεριφέρονται οι καταναλωτές. Τους ρωτούμε λοιπόν πόσο συχνά αντιμετωπίζετε προβλήματα με συγκεκριμένα αγαθά, ε, με ελαττωματικά αγαθά και όταν προκύπτουν αυτά τα ελαττώματα, ε, τι συμβαίνει. Και τι διαπιστώσαμε. Ε, κατά μέσο όρο, 96% των προβλημάτων προκύπτουν πριν πριν ολοκληρωθεί η διετής εγγύηση και μεγάλος αριθμός ε, των προβλημάτων προκύπτουν τους πρώτους μήνες της χρήσης. Επίσης σημαντικό είναι να γνωρίζουμε, βεβαίω ε, μιλήσαμε κυρίως με καταναλωτές ε, στη Σουηδία, στην Ολλανδία, στην Φιλανδία όπου η περίοδος, η περίοδος εγγύησης είναι μεγαλύτερη και στις χώρες εκείνες πάντως οι καταναλωτές μας λένε ότι το ποσοστό των ελαττωμάτων που εμφανίζονται μετά τα δύο χρόνια είναι πολύ μικρό. 2% στη Σουηδία έως 7% ε, maximum στην Φιλανδία. Σημαντικό είναι να διαπιστώσουμε ότι στις χώρες αυτές οι κατηνοδετές ε, δεν γνωρίζουν επαρκώς τα δικαιώματά τους. Ε, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ε, ενώ η οδηγία αυτή υπάρχει 20 χρόνια τώρα. Οι καταναλωτέ, σε χώρες όπου υπάρχει μια πολύ πιο γενναιόδορη γενναιόδορη καθεστώς σε επίπεδο δεν τα γνωρίζουν αυτά. Πολλοί μας λένε παραδείγματος χάρη ότι έχουν δύο χρόνια εγγύηση, έτσι νομίζουν, είναι παραπάνω. Να περάσουμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια. Show us. Εδώ βλέπουμε τι πιστεύουν οι επιχειρήσεις. Τι πιστεύουν ότι θα ήταν το κόστος και το όφελος από μια πιθανή εναρμόνιση της νόμιμης περιοδογγίσης των δύο ετών. Λοιπόν, το 13% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι μια τέτοια πιθανή εναρμόνιση θα μειώσει το κόστος σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Εσείς μπορεί να ισχυριστείτε ότι δεν είναι τεράστιο το ποσοστό, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι αυξάνεται εάν ρωτήσουμε τους επιχειρηματίες της Σουηδίας, της Φιλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των κάτω χωρών σε λιγότερο βαθμό. Είναι λοιπόν ένας τομέας αυτός όπου ε, βλέπουμε από τους ενδιαφερομένους ότι οι επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται υπό το παρόν καθεστώς θεωρούν ότι θα ήταν πολύ καλύτερο ένα ομοιόμορφο, σαφέ κανονιστικό καθεστώ ε, το ίδιο σε ολόκληρη την Ευρώπη και πιστεύουμε ότι πολύ πιθανόν αυτό να εξοικονομήσει και κόστη. Α περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια όπου θα δούμε ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο πολιτική, την επιλογή του κατά πόσο πρέπει να αντιστρέψουμε το βάρο τη απόδειξη. Εδώ έχουμε την ερώτηση που κάναμε στους επιχειρηματίες από τους οποίους θέλαμε να μάθουμε αν η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης κατά δύο έτη θα είχε κάποια επιρροή πάνω σε αυτούς ε, από αψικούς τους και ωφέλους. Το ενδιαφέρον που μάθαμε είναι ότι πολλές επιχειρήσεις και μάλιστα είναι αυξανόμενος ο αριθμός ε, όσο συνεχίζει η ανάλυση από τον αναδοχό μας ε, και όπως συνέχισε μέσα στον Αύγουστο με όλο και περισσότερες ερωτήσεις επιχειρήσεις. Πολλές λοιπόν επιχειρήσεις λένε ότι κάτι τέτοιο θα είχε ελάχιστες επιπτώσεις στο κόστος ή καθόλου. Οι επιχειρήσεις λοιπόν είναι διατεθειμένες να θεωρήσουν ότι αυτός είναι ένας καλός κανόνας διότι θεωρούν ότι ο κανόνας αυτός θα περιορίσει και το κόστος των διαφορών και της επίλυσης των παραπονών και των διαφορών. Μια μελέτη του 2015 για τα ε, νομικές και ε, εμπορικές ε, εγγυήσεις που δημοσιεύθηκε πριν από λίγο καιρό έδειξε ότι οι λιανοπολιτές είναι ιδιαίτερα ευγενικοί προς τους πελάτες. Δεν αρχίζουν να λένε «Α, το αγοράσετε πριν από 6-7-18 μήνες». Απλά προσπαθούν να βρουν μια λύση στη μία περίπτωση ή είναι εχθρικοί προς τους πελάτες και μετράνε την κάθε μέρα. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει κάποια ευελιξία στον τομέα αυτόν κάτι φυσικά εξαιρετικά σημαντικό από την άποψη των καταναλωτών, ε, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της άσκησης των δικαιωμάτων τους. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε την ιεραρχία των ένδικων μέσων. Από τα πρώτα δεδομένα που έχουμε συλλέξει βλέπουμε κάτι γνωστό από την καθημερινότητα. Το 51% των καταναλωτών είτε δεν ζητούν άμεση έκπτωση ή λήξη τη σύμβαση ε, ή το κάνουν μόνο αν δεν επιληθεί το πρόβλημα μετά από την πρώτη επισκευή ή αντικατάσταση. Δεν είναι λοιπόν συντριπτική πλειοψηφία, αλλά είναι μια πλειοψηφία καταναλωτών που απλά δεν το πράττουν. Θεωρούν ότι είναι λογικό να δώσουν μια δυνατότητα στον πολιτή να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν. Ακόμη και σε χώρε όπω η Κροατία, η Λιθουανία και η Ελλάδα, όπου υπάρχει νομική ελεύθερη επιλογή ένδικων μέσων, αντίστοιχα 67%, 60% και 50% των καταναλωτών δεν ζητούν άμεσα έκπτωση ή λήξη της σύμβασης. Η μελέτη του 2015 για τις νομικές και εμπορικές εγγυήσεις μας έδειξε και άλλα ενδιαφέροντα γεγονότα. Όταν ε, ρωτήθηκαν άμεσα, το 77% των καταναλωτών συμφώνησαν ότι είναι πολύ λογικό ένας πολιτής να προσφέρει πρώτα επισκευή ή αντικατάσταση σε περίπτωση προβλήματος ε, κατά την πρώτη χρήση ενός προϊόντος. Και αυτό πιστεύω πρέπει να ληφθεί υπόψη. Στην επόμενη διαφάνεια θα σας πω τα τελευταία μου λόγια για την τελευταία ε, επιλογή πολιτικής. Πρόκειται για άλλο ένα κανόνα που προτείναμε ήδη από το Δεκέμβριο για την άρση μιας υποχρέωσης προς τον καταναλωτή να κοινοποιεί το ελάττωμα εντός δύο μηνών αφού το ανακαλύψει. Εδώ ανακαλύψαμε το εξής. Το 62% των επιχειρήσεων και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πω ότι συνεχίζει να αυξάνεται το νούμερο καθώς προχωράει η ανάλυση του αναδόχου μας αυτοί λοιπόν θεωρούν ότι η άρση μιας τέτοιας υποχρέωσης κοινοποίησης δεν θα ε, συνεπάγεται κανένα κόστος ή ελάχιστο κόστος. Έχουμε επίσης στοιχεία που δείχνουν ότι σε γενικές γραμμές οι καταναλωτές ε, όταν εντοπίσουν κάποιο πρόβλημα κάνουν κάτι γι' αυτό. Ανάλογα με το προϊόν, μεταξύ 37% και 58% αυτών κάνουν αμέσως κάτι, ειδοποιούν αμέσως τον πολιτή ή εντός μιας εβδομάδας. Δηλαδή, όπω φαίνεται, συνήθω ε, προσπαθούν να δείξουν κάποια λογική συμπεριφορά οι καταναλωτέ και πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο χρειαζόμαστε κάποια τέτοια διαδικασία. Με μεγάλη μα χαρά θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εδώ είμαστε μόλι στην αρχή τη όλη διαδικασία, όπω είδατε. Και φυσικά και εγώ και οι συναδελφοί μου είμαστε στη διάθεσή σα για να απαντήσουμε σε ερωτήσει. Ευχαριστώ. Thank you, Vicky. Ευχαριστώ, Βίκη. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Κομισιόν που μας παρουσίασε τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία επίσης μας δίνουν ε, σημαντικά συμπεράσματα. Θα ήθελα όμως να προστάσω ότι, προς, πρόκειται για κάποια πρώτα, ε, ε, για πρώτα στοιχεία, τα οποία όμως θα πρέπει να εξετάσουμε λεπτομερέστερα, όπως είναι για παράδειγμα ο ρυθμός των καταναλωτών ε, που εξετάστηκαν, ναι, είναι καλός αριθμός, όμως αναρωτιέμαι αν οι 375 ε, επιχειρήσεις που ερωτήθηκαν, αν αυτό αποτελεί μια υγιή ισορροπία σε σχέση με τον αριθμό των ε, καταναλωτών που ερωτήθηκαν. Αυτό ίσως θα πρέπει να αυξηθεί με αποτέλεσμα κατά συνέπεια να αναπροσαρμοστούν και τα δεδομένα. Τώρα όσον αφορά τα πρώτα συμπεράσματα ε, και σχόλια τα οποία μπορώ να βγάλω εγώ είναι το γεγονός ότι φαίνεται ε, πως ε, οι έμποροι, τα υπουργεία, οι κυβερνήσεις υποστηρίζουν ε, η online και η offline αγορά ε, να ενωθούν ε, το 37% των εμπόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν και επικοινωνικές πωλήσει και θεωρώ ότι συνεχίζει να αυξάνεται το συγκεκριμένο φαινόμενο. Επίσης θεωρώ ότι δεν υπάρχει μία και μόνο απόδειξη εδώ πέρα σχετικά ε, με την ε, νόμιμη εγγύηση των δύο ετών να αυξηθεί αυτή δεν νομίζω ότι το υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Στη Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία, κάτω χώρε Φινλανδία και Σουηδία υπάρχει μεγαλύτερη περίοδος, όμως δεν θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο. Οι καταναλωτές ε, θεωρούν ότι τα δύο έτη επαρκούν, κάτι το οποίο βρίσκω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον ως παρατήρηση. Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε ότι ε, η σύνδεση της εγγύησης με την ε, διάρκεια ζωής των συγκεκριμένων προϊόντων ε, θα είναι αρκετά πολύπλοκο διότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα τα χρησιμοποιούν καθημερινά θεωρούν ότι κάτι τέτοιο θα τους είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Τώρα όσον αφορά την ε, υποχρέωση της απόδειξης, ε, το 69% των περιπτώσεων ε, δείχνει ότι οι καταναλωτές, οι περισσότεροι καταναλωτές συνειδητοποίησαν το πρόβλημα εντός της περίοδου της εγγύηση, ενώ το 45% μάλιστα την πρώτη και όλες εβδομάδα. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη μας όσον αφορά την ιεραρχία. Το 77% των καταναλωτών το υποστηρίζουν και έρχεται σε αντίθεση με το γεγονό ότι στο 45% των καταναλωτών τα στοιχεία αυτά ε, θέλουν ε, να, διακόψουν ε, την συνδρομή, την, θέλουν τα χρήματα τους πίσω σε περίπτωση που αποδειχθεί κάποιο πρόβλημα. Και όσον αφορά τα συμπεράσματα, θα πρέπει να μάθουμε περισσότερα και για τα ερωτήματα. Ίσως θα πρέπει να ενημερωθούμε για αυτά σε, μια επόμενη συνάντηση για να μπορέσουμε να αναλύσουμε το τη σχέση που έχει το ερώτημα με, το, με τα δεδομένα. Σύμφωνα με τον πίνακα 1,3 δεν υπάρχει, ε, υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο δεν αγοράζει ποτέ εκτός συνόρων, το οποίο αποτελεί έκπληξη. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν τα δεδομένα αυτά φορούν ε, καταναλωτές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα χρόνων στην, στον πίνακα 2,5 ε, επιβεβαιώνεται κάτι το οποίο φαίνεται και στον πίνακα 2,7 και 2,8 ότι, ότι μια υψηλότερη προστασία των καταναλωτών δεν θα οδηγήσει και σε επιπρόσθετα κόστη. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω ακριβώς το ερώτημα το οποίο ετέθη στους ε, εμπόρους ε, διότι σε 375 επιχειρήσεις θα ήθελα να δω δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται όλε οι επιχειρήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύπτονται με 375 επιχειρήσει που ερωτήθηκαν. Και θα ήθελα να απευθύνω και κάποια ερωτήματα προ την Κομισιόν. Το πρώτο είναι πώς εσείς υποστηρίζετε την σύνδεση του online και, του, και των offline αγορών. Το δεύτερο αφορά ε, όταν μιλάμε για, τις, ε, για την νόμιμη εγγύηση, τι υποστηρίζει να τις αυξήσουμε ή το κάνουμε αυτό απλά και μόνο για να ικανοποιήσουμε τον καταναλωτή και πώς σκέφτεται να συνδέσει την εγγύηση με το βιώσιμο των προϊόντων και το τρίτο μου ερώτημα αφορά την ε, ιεραρχία των ένδικων μέσων η ε, Κομισιόν ε, θεωρεί ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός αυτών οι οποίοι υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Είναι υπέρ και ε, ανυπομονώ να ακούσω τις απαντήσεις σας. Lucy Anderson. Ευχαριστώ εμείς ε, από το S&D, από τους δημοκράτες, ε, χαιρόμαστε για την έρευνα αυτή της Κομισιόν. Έχουμε και εμείς όμως κάποιες ανησυχίες, όπως είπε και ο κύριος Άραμον, για τη μεθοδολογία που ακολουθείτε. Ποια ερωτήματα θέτετε έτσι. Είναι σημαντικό αυτό, διότι είναι διαφορετικό. Ε, έχει μεγάλη διαφορά μάλλον ανάλογα με το ποιο αγαθό μιλάμε. Το ερώτημα, παραδείγματος χάρη για τις νομικές εγγυήσεις, δείχνει ότι 34-43% των ε, απαντήσεων θεωρούν τα δύο χρόνια είναι επαρκή. Ε, για τις ε, ε συσκευές, τις συσκευές. Αλλά γιατί συσκευές μιλάμε. Ε, μια ένωση καταναλωτών στη χώρα μας έχει αποδείξει ότι δεν χαλάνε οι κοσκευέ, πολλές τα δύο πρώτα χρόνια, αλλά χαλάνε, χαλάνε αμέσως μετά. Το να έχουμε λοιπόν μια εγγύηση πάνω από, δύο χρόνια, πάνω από δύο χρόνια είναι ένα σημαντικό θέμα ε, και δεν πρέπει έτσι ελαφρά την καρδία να το ε, αποκλείσουμε. Με ενσυχεί κάπω γενικά και σε παιδονομικό και σε παιδοδικαιωμάτων του καταναλωτή αυτό που γίνεται. Οι καταναλωτέ αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να εφαρμόσουν, ε, να ασκήσουν τα δικαιώματα τα οποία τους αντιστοιχούν. Δεν μπορούμε εδώ να έχουμε ένα παζάρι μεταξύ χωρών και τελικά να, αυτό να είναι εις των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Είναι υποκειμενικά τα ερωτήματα αυτά. Από νομική πλευρά πρέπει να δούμε όμω αντικειμενικά το θέμα των δικαιωμάτων του καταναλωτή με βάση το δίκαιο και τη δικαιοσύνη και όχι με το τι θεωρεί ο τάδε ο δίνα ως λογικό. Ε, οι ερωτήσεις λοιπόν αυτές κάπως τον προβληματίζουν. Επίσης δεν ξέρω αν τέθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα για το βραχυπρόθεσμο δικαίωμα απόρριψης. Βλέπω σε κάποια αποτελέσματα ότι οι καταναλωτέ σε γενικές γραμμές ε, ε, συνήθως δεν καθυστερούν. Όταν δηλαδή προκύπτει κάποιο πρόβλημα το θέτουν αμέσως όταν υπάρχει κάποιο ελάττωμα. Το δικό μας νόμο, ε, γι' αυτό έχουμε ένα μικρό χρονικό διάστημα αντίδρασης. Μπορεί κάποιος δηλαδή, εφόσον ε, αντιδράσει έγκαιρα, να στείλει πίσω το, το προϊόν. Είναι βασική αρχή αυτή. Και η έρευνα σε κάποιο βαθμό το υποστηρίζει αυτό. Χαίρομαι λοιπόν για την έρευνα αυτή, αλλά νομίζω ότι θέτει πιο πολλά ερωτήματα από ότι απαντήσεις. Ευχαριστώ Βίκη να μιλήσω εκ μέρους της Ανελή που δεν βρίσκεται εδώ σήμερα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστεί την Κομισιόν για την παρουσίαση της άσκησης REFIT. Στο πλαίσιο της βελτίωσης της νομοθεσίας η Ανελής ανέκαθεν υποστήριζε να περιμένουμε το REFIT πριν ξεκινήσουμε ε, τις, ε, ε, την εργασία και τις κλασικές πωλήσει και τις online πωλήσει. και χαιρόμαστε τώρα που γνωρίζουμε κάποια περισσότερα πράγματα για το Refit και μπορούμε να προχωρήσουμε με τις εργασίες μας. Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο θα επεκτείνουμε το αντικείμενο της πρότασης για τις offline και τις κλασικές πωλήσει και όπως δείχνει η μελέτη είναι απαραίτητο. Είμαστε σε μια εποχή όπου παλιά οι πελάτες αγόραζαν στα καταστήματα και σήμερα όλο και περισσότερο στο διαδίκτυο και πρέπει να χαιρούν κάποιου επαρκούς επίπεδου προστασίας ανεξάρτητα από τον τρόπο. Και εμάς, ως νομοθέτης έχουμε το καθήκον να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα για αυτούς. Επίσης και για τους λιανοπολιτές όταν ε, ε, κάνουν και τους δύο τύπους πωλήσεων πρέπει και για αυτούς τα πράγματα να είναι πιο σαφή. Όπως επισημαίνουμε στην εκθέση το 35% των ε, λιανοπολιτών στην Ευρώπη πράττουν και τους δύο τύπους πωλήσεων και ξέρετε, στην Ευρώπη μια μεγάλη πλειοψηφία είναι πολύ μικροί λιανοπολιτέ. Το γεγονό ότι το 35% ε, είναι πλέον το ποσοστό αποτελεί έδειξη ότι όλο και περισσότερο οι online πωλήσει ε, θα χαρακτηρίζουν τι αγορέ στο μέλλον στην Ευρώπη. Ε, από την πλευρά των συντονιστών, από όσον αφορά τα δύο έτη και τα γενικά δικαιώματα των καταναλωτών όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή, πρέπει να μην αποδυναμώσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών όπως υπάρχουν στα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή. Και όπως επισήμαναν και οι προηγούμενοι ομιλητές σε πολλά κράτη-μέλη, ε, η νομοθεσία των δικαιώματων των καταναλωτών είναι ισχυρότερη από ό,τι προτείνουμε εδώ, οπότε πρέπει να μην αποδυναμωθεί αυτή η νομοθεσία, γιατί δεν θα αρέσει αυτό καθόλου στου καταναλωτέ. Και κάτι άλλο που ανέφερε και η Λούση Άντερσον, ακόμη και αυτή τη στιγμή οι καταναλωτέ δεν γνωρίζουν απόλυτα τα δικαιώματά του. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε, να προσέξουμε αξιοποιώντα τα αποτελέσματα ερευνών, διότι συχνά οι καταναλωτέ δεν γνωρίζουν όλα του τα δικαιώματα. Οπότε πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να τα γνωρίζουν καλύτερα. Τώρα γενικά οι αναλύση ε, είναι ικανοποιημένοι με τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα του Refit ε, και αυτό επιβεβαιώνει τη σύσταση που είχαν κάνει τότε οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι και προσβλέπει στο να Συνεχίζει τη μελέτη των αποτελεσμάτων αυτή, αυτών με τον εισηγητή και τους συνεισηγητές και τους κοιόδης ε, ώστε να βελτιστοποιηθεί αυτή η πρόταση στο μέλλον. Ευχαριστώ. Καία Καλάς. Sorry, been away. Κατανοώ ότι τα συμπεράσματα του ε, Ρεφίτ ε, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ε, και τις ε, offline πωλήσει, όμως το ερώτημα το οποίο γίνεται είναι αν αυτό το καθεστώς τόσο για τις συμβατικές πωλήσει όσο και τις εξαποστάσεως απαιτείται και αν υπάρχουν απαντήσεις που λένε ότι σε ένα νομοθετικό καθεστώς θα υπάρχει διαφοροποίηση για συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία ίσως να προκύψουν σε περίπτωση που υπάρχει μία offline ή online πώληση. Αλλά αν δεν υπάρξει διαφοροποίηση των ε, πωλήσεων, τότε ίσως θα πρέπει να αντιμετωπίζετε το ίδιο. Υπάρχουν ακόμα διαφορές και το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο φαινόμενο. Στους σκιώδεις έχω Πασκάλ τεγόν. Όμως πρώτα θα μιλήσει η Τζούλια Ρέιντας, κάποιος άλλος από τους κοιόδης. Αρχικά λοιπόν η Τζούλια από τους Πράσινους. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, τα οποία θεωρώ είναι ε, σημαντικά ε, για το έργο που κάνουμε. Πιστεύω ότι θα πρέπει λοιπόν να στοχεύσουμε σε μια συνοχή μεταξύ των κανονισμών για τις offline και online πωλήσει. Όμως δεν μου είναι ξεκάθαρο σε ορισμένα σημεία ε, τα, τι συμπεράσματα βγάζει η Κομισιόν και το πώς θα τα επεξεργαστεί αυτά συγκεκριμένα όσον αφορά την ελεύθερη επιλογή για τα ένδικα μέσα όπως ε, γνωρίζουμε από τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάστηκαν, έχουμε την ιεραρχία των μέσων. Υπάρχουν ε, κάποια κρατημέλη τα οποία έχουν ελευθερία σε αυτό το ζήτημα και αν καταλαβαίνω καλά την Κομισιόν προτείνεται να αφαιρέσουμε αυτή την ελεύθερη επιλογή και να εφαρμόσουμε μια ιεραρχία ενδικών μέσων σε όλες τις περιπτώσεις. Ε, δεν βλέπω να υποστηρίζεται αυτό με τα συγκεκριμένα δεδομένα. Έχετε μία αναφορά όπου αρκετοί καταναλωτές έχουν την ελεύθερη επιλογή και κάνουν χρήση αυτής. Ε, βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής πάντοτε θα επιλέγει ε, να ζητά πίσω τα χρήματά του. Όμως ανάλογα με το αγαθό η επιστροφή χρημάτων μπορεί να είναι πιο χρήσιμη ή όχι, όμως ε, συγκεκριμένα όσον αφορά τον τομέα των ψηφιακών αγορών, μια τάση την οποία παρατηρούμε είναι ότι υπάρχουν ε, πολλές ε, αγορές από μικρά καταστήματα με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται όλο και πιο ελκυστικό, όπως για παράδειγμα να πουληθεί ένα MP3 για 50 cent και σε αυτή την περίπτωση, περίπτωση να περάσει μια τέτοια ιεραρχία όταν δεν έχεις λάβει αυτό ε, που έλαβες, ε, που πλήρωσες, τότε το να ζητήσεις πίσω τα χρήματά σου δεν φαίνεται πολύ λογικό. Επίσης, πολλοί καταναλωτές λαμβάνουν δράση σε περίπτωση ε, που υπάρχει ένα προβληματικό αγαθό. Το 90% το κάνει αυτό είτε έχει την επιλογή είτε όχι και φυσικά φυσικά δεν αποτελεί έκπληξη διότι οι περισσότεροι καταναλωτές σίγουρα θα κάνουν κάτι σε περίπτωση που δεν λάβουν αυτό το οποίο περίμεναν και θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα που τους είναι διαθέσιμα δεν βλέπω όμως κάποια δεδομένα τα οποία να δικαιολογούν ότι δεν είναι αναγκαία η ελεύθερη επιλογή ενδικών μέσων. Οπότε θεωρώ ότι εν τέλει είναι μια πολιτική απόφαση. Θα ήθελα να μάθω από την Κομισιόν με βάση τα αποτελέσματα του Ράφιτ και με βάση τις απαντήσεις αν θα προτείνατε κάποιες αλλαγές στις προτάσεις που μας παρουσιάζεται το Δεκέμβριο Αναφέρθηκε ήδη το ζήτημα σχετικά με το αν θα επεκταθεί ε, το ε, εύρος για τα ε, συμβατικά προϊόντα τα οποία πολλούνται. Έχει, έχουν υπάρξει κριτικά, επικριτικά σχόλια και ερωτήματα σχετικά με το αν θα παρουσιαστούν πριν από το REFIT. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω αν το REFIT άλλαξε την, τον τρόπο που το αντιμετωπίζετε. Λοιπόν, η Evelyn Gebhardt πρώτα, αλλά πριν θέλω να χαιρετήσω μια ομάδα από τον Νόι Ούλμ που βρίσκεται εδώ πίσω στην αίθουσα και μας παρακολουθεί. Υπάρχει νομίζω και υπάρχουν εδώ και εκπρόσωποι ε, των ε, δημοσίων υπηρεσιών του Μπράντεμπουργκ. Εμείς πάντα καλωσορίζουμε τους πολίτες στην ομάδα μας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Είναι με πολύ σημαντική επιτροπή. Εξετάζουμε ζητήματα προστασία των καταναλωτών, δικαιωμάτων των καταναλωτών που να αγοράζει κάποιο επιγραμμικά προϊόντα και η Evelyn Gebhardt ε, είναι ένα θέμα που την συναρπάζει ε, και την παθιάζει και ελπίζω να βλέπετε με πόσε πώς λεπτομέρειε εξετάζουμε σχετική νομοθεσία. Evelyn, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Βίκη. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερως όταν έχουμε επισκέπτες ανάμεσά μας, ώστε να παρακολουθήσουν τι δουλειά κάνουμε εμείς οι ευρωβουλευτές και το πώς ε, συνεργαζόμαστε για ζητήματα τα οποία ξεπερνούν τα σύνορα. Το θέμα λοιπόν το οποίο μας αποσχολεί σήμερα είναι σημαντικό και θα ήθελα να συμφωνήσω ε, με τον συνάδελφο θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ερωτήθηκαν, αν υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ των ε, συνοριακών περιοχών όπου ε, είναι πιο σύνηθες να αγοράζουν ε, σε γειτονικέ χώρες για παράδειγμα, όταν κοιτάζω την Βιδεμβέργη, η κατάσταση θα είναι διαφορετική από ότι σε άλλες περιοχές. Το δεύτερο ζήτημα δείχνει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλοί καταναλωτές δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε λεπτομερέστερα. Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να επιληθεί με το Refit, όμως θα επηρεάσει σίγουρα τις απαντήσεις των πολιτών. Γι' αυτό και θα πρέπει να το εξετάσουμε. Και το τρίτο το οποίο θα ήθελα να μάθω είναι αν θα μπορούσαμε να έχουμε ολόκληρο τον κατάλογο των ερωτημάτων έτσι όπως τέθηκε, διότι ο τρόπος με τον οποίο τίθενται τα ερωτήματα είναι σημαντικός για να μπορέσουμε να καταλάβουμε σχετικά με τις απαντήσεις που δίνονται και αποτελούν και μία ένδειξη σχετικά με το αν ε, οι απαντήσεις που δίνονται ήταν σωστές ή λάθος. Όσον αφορά την ιεραρχία των ένδικων μέσων, παρατηρώ στον πίνακα ότι δεν γνωρίζουν ε, ότι οι εναλλακτικές είναι δεν γνωρίζω, free choice, ελεύθερη επιλογή, ε, αυτό μπορεί να μπερδέψει τους καταναλωτές λοιπόν, διότι εκεί υπάρχει διάκριση μεταξύ του αν είναι ελεύθερο ή αν έχουμε μια κατευθυντήριο σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Υπάρχει λοιπόν μια διαφοροποίηση. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πώς ακριβώς έχουν τεθεί τα συγκεκριμένα ερωτήματα για να μπορέσω να αξιολογήσω καλύτερα το πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τα συγκεκριμένα στατιστικά αποτελέσματα. Θα ήθελα περαιτέρω ε, λεπτομέρειες, κάτι το οποίο μας παρουσιάσατε και στην παρουσίασή σας, ότι όσον αφορά τις επιχειρήσεις δεν είναι εν τέλει από οικονομικής άποψης ε, δεν τους αφορά ιδιαίτερος λοιπόν εάν η εγγύηση θα είναι δύο χρόνια ή και περισσότερο ε, συμφωνώ με όλους σήμερα ότι κανένας καταναλωτής θα πρέπει να χάσει δικαιώματα από μια εναρμόνιση της νομοθεσίας. Ξέρουμε ότι τα δικαιώματα είναι διαφορετικά και εγγυήσει τριών χρόνων στη Γαλλία, έξι ε, σε περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας, ε, Μεγάλης Βρετανίας, μόλις δύο χρόνια στη Γερμανία. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν να στο κάνουμε όλοι δύο χρόνια αυτό ε, δεν μας ενδιαφέρει διότι πολύ απλά οι Μεγάλοι Βρετανοί δεν, οι Βρετανοί δεν γνωρίζουν ποιο είναι το νόμιμο, η νόμιμη εγγύηση. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για εμάς και γι' αυτό το λόγο χρειάζομαι και άλλες πληροφορίες για να μπορέσω να καταλάβω καλύτερα τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο κύριος Γκουόγκα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δημιουργείται μια κάποια σύγχυση. Ε, είναι σωστό αυτό που ελέγχθη, ότι δεν έφτασαν υπαρκώς υπόψη οι επιχειρηματίες στην έρευνα. Των μικρών επιχειρήσεων εκπρόσωποι μπορεί να μας δώσουν μια σαφέστερη ένδειξη. Αυτό ίσως να δείχνει ότι δεν ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση Έγινε γρήγορα η εξολόγηση αντικτύπου, ε, βιαστικά και η έρευνα αυτή μάλλον θα κάνει πιο πολύ κακό παρά καλό στην ενιαία αγορά. Θέλουμε ενιαία αγορά, έτσι, ε, και επιγραμμικά και μη επιγραμμικά. Αυτό είναι ο στόχο μα. Μην ξεχνάμε αυτό το στόχο. Και εμεί πιστεύουμε ότι αυτό πάει προ τη λάθο κατεύθυνση. Η Κομισιόν, κατά τη γνώμη μα, πρέπει να αποσύρει την πρόταση και να υποβάλει μια νέα πρόταση και για επιγραμμική και για μη επιγραμμική πώληση με ε, μέγιστη εναρμόνιση. Οι κανόνες ε, που αντι, αντίκυνται στην ε, εναρμόνιση είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια στο διασυνοριακό εμπόριο. Ναι, ξέρω ότι πρέπει να πάτε και σε μια άλλη συνεδρίαση. Σκοπεύετε να το δημοσιεύσετε αυτό ε, θα το δημοσιοποιήσετε, θα το συμπεριλάβετε δηλαδή στη διαβούλευση. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να δούμε βεβαίως τα ερωτήματα που θέτετε, διότι οι καταναλωτές επίσης μπορούν να αντιδράσουν διαφορετικά ανάλογα με το αγαθό. Λέτε, παραδείγματος χάρη, ρωτάτε, ε, αντιδράσατε, διαμαρτυρηθήκατε απευθεία στον πολιτή. Εγώ έχω την τάση ε, να διαμαρτυρηθώ και να αντιδράσω αν είναι υψηλότερη αξία το αγαθό. Δηλαδή το γεγονό ότι οι πολίτε δεν ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά του δεν σημαίνει πρέπει να τα πάρουμε κιόλα. Ε, το δικαίωμα επιστροφή στη χώρα μου είναι ένα δικαίωμα το οποίο το γνωρίζουν καλά οι συμπολίτε μα αλλά δεν καλύπτονται. Αλλά δεν καλύπτεται εδώ και κάτι για τι επισκευέ. Οι καταναλωτέ ε, δεν του αρέσει το δικαίωμα στην επισκευή και ξανά επισκευή, ξανά επισκευή, ναι το έφτιαξα, όχι δεν, ναι, δεν, το, δεν το έφτιαξες, δεν είναι πάντα ότι καλύτερο. Θέλετε να απαντήσετε κάποια τα ερωτήματα, ίσως να χρειαστούμε πάντως και γραπτός κάποια περαιτέρω στοιχεία. Thank you, Chair. Thanks. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλα τα αξιότιμα μέλη που πήραν το λόγο. Να επαναλάβω πρώτα απ' όλα αυτό που αναφέρεται και στην επιστολή της Κομισιόν. Λαμβάνεται ουσιαστικά ένα ερωκτικό εδώ. Αρχικά στοιχεία λίγο επεξεργασμένα. Τέλη Σεπτεμβρίου θα έχετε την τελική έκθεση με όλα αυτά τα στοιχεία που σχετίζονται με την ευθυγράμμιση των κανόνων για τις offline και τις ε, online ε, πωλήσει. Ναι, θα υπάρξει μια τελική έκθεση η οποία θα δημοσιευτεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα αυτή τη στιγμή είναι ένας ειλικρινής δημοσιολογητής σε μια νομοθετική διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει και προσπαθούμε να σας ε, παρέχουμε τα καλύτερα μας πορίσματα, ευρήματα που σχετίζονται με το τι έχουμε πετύχει. Εγώ πρώτη απ' όλα έχω απογοητευτεί που επικοινωνήσαμε μόλις με 375 επιχειρηματίες αντί για 500, όπως είπε ο εισηγητής ο κ. Σαρημών. Μπορείτε εσείς να μας βοηθήσετε να βελτιωθούμε. Δημοσιεύσαμε μια δημόσια διαβούλευση online για το REFIT ε, εδώ και πάνω από 12 εβδομάδες και έχουμε λάβει μόνο 300 απαντήσεις. Θέλω να με βοηθήσει η Επιτροπή σας να μιλήσουμε με περισσότερους πραγματικούς καταναλωτές, με περισσότερες επιχειρήσεις. Είναι σημαντική η επαφή με όλους αυτούς και πρέπει να το κάνουμε ενωμένα. Αλλά σας εγγυώμαι ότι εδώ αυτοί που απάντησαν είναι πραγματικοί επιχειρηματίες και μικροί επιχειρηματίε και μεσαίοι. Πολλές φορές ακούμε πολλά από τις μεγάλε επιχειρήσει ή οργανισμού ε, με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα χωρίς ε, τοπική εμπειρία και αυτοί έχουν κάποια εμπειρία, αλλά εντάξει, να ξέρετε, πάντα θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα, πάντα θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Όσον αφορά τους καταναλωτές, με μεγάλη μας χαρά να σας παράσχουμε τις πληροφορίες από αυτό το αντιπροσωπευτικό δείγμα όλων των ηλικιών και κοινωνικών προελεύσεων. Οπότε δεν θα υπάρχει ε, πρόβλημα, θα υπάρχει δυνατότητα να δείτε ε, τους τόπους κατοικιών των ανθρώπων ε, που ερωτήθηκαν στα 28 κρατημέλη καθώς και στην Ισλανδία και την Νορβηγία. Επίσης με μεγάλη μας χαρά να σας κοινοποιήσουμε και το ερωτηματολόγιο. Σύμφωνα απόλυτα με τα σχόλια πολλών ομιλητών ότι ορισμένα από τα προαρτήματα θα γίνουν πιο κατανοητά όταν ε, θα βάλει κάποιος δίπλα και τα ερωτήματα. Οπότε ευχαριστώ να σας δώσουμε και τις ερωτήσεις. θα κλείσω εδώ, γιατί όπως είπα δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε φάση που να μπορούμε να ε, ισχυριζόμαστε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές. Διατηρώ τη θέση που προτείναμε το Δεκέμβριο. Αυτό που προτείναμε το Δεκέμβριο εξακολουθεί να είναι μια εύλογη προσέγγιση. Κανένα από τα στοιχεία που σας παρουσιάζουμε δεν έρχεται σε αντίθεση με το εύλογο αυτής της προσέγγισης, αλλά φυσικά υπάρχει περιθώριο να συζητήσουμε τις διάφορες επιλογές να δώσω το λόγο στον Τύρξ Τεδεμάιερ για τον συναδελφό μου για κάποιε περαιτέρω παρατηρήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να απαντήσω σε ορισμένα από τα σχόλια του εισηγητή κυρίου Άριμον και της κυρίας Ρέντα και δικά σας ε, σχόλια που κάνετε στο τέλος σε σχέση με την πρόταση. Ο κύριος θα ήθελα να ρωτήσω, ε, ρωτήθηκα ε, σχετικά με την άποψη για τις online πωλήσει. Υπόθηκε η πρόταση ότι είναι σημαντικό τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις να έχουν ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν όποτε ε, αγοράζουν και πολλούν online ή offline. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι τα δεδομένα τα οποία έχουμε και τα οποία έχουμε εξετάσει επιβεβαιώνουν τη συγκεκριμένη άποψη. Όπως είπε η Βερόνικα, η ιδέα, μου, η ιδέα μας είναι να ε, συμπεριλάβουμε τα συγκεκριμένα δεδομένα στην νομοθετική διαδικασία τόσο για εσάς όσο και για το ε, Συμβούλιο και να μπορέσουμε να επεκτείνουμε το πλαίσιο δράσης. Δεύτερον, ρωτήσατε για το ζήτημα της εγγύησης ε, των δύο χρόνων ή αν θα πρέπει να συνδεθεί με το βιώσιμο του προϊόντος. Η Κομισιόν ε, πρότεινε ε, μια διετή εγγύηση για διάφορους λόγους, τους οποίους όμως δεν θα αναφέρω όλους. Θα ήθελα όμως να αναφέρω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους προτείναμε το συγκεκριμένο μοντέλο είναι ότι ε, θα διασφαλίζει τη δικαιοσύνη διότι ισχύει για όλους, για όλα τα κράτη-μέλη και έτσι λοιπόν είναι πιο εύκολο να ε, γίνονται πωλήσει online και offline. Επίσης, ε, ακούσαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές εγγυήσεις από διάφορα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν αν πρέπει κατά περίπτωση να αποφασίσουμε ποια εγγύηση ισχύει, τότε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές κατάστασεις και όχι στην ε, διασφάλιση του δικαίου. Τώρα ως μια απάντηση στην κυρία Για ποιο λόγο μέσω της, ε, θα πρέπει να ακολουθήσουμε την ιεραρχία η διαφορά αυτής της ε, πρότασης σε σχέση με την οδηγία του 1999 είναι ότι η μετάβαση από την πρώτη στη δεύτερη βαθμίδα γίνεται πιο εύκολη και αυτό περιλαμβάνεται στις προϋποθέσεις ε, σύμφωνα με το άρθρο 9 είναι λοιπόν εμφανώς πιο εύκολο να λήξει ένα συμβόλαιο για παράδειγμα και δεν είναι αναγκαίο έτσι λοιπόν σε όλες τις περιπτώσεις να ε, εφαρμόζονται όλες οι διαδικασίες. Και τέλος, κυρία Φόρτ, ε, κάτι τελευταίο το οποίο ρωτήσατε όσον αφορά τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες επισκευής. Ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει να αποφύγει η Κομισιόν και γι' αυτό το λόγο έχουμε τονίσει ε, στο σημείο 58 της πρότασης ότι ε, ο καταναλωτής ε, δεν θα πρέπει να υπόκειται σε επαναλαμβανόμενες προσπάθειες επισκευών. Θα πρέπει να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο θα πρέπει το προϊόν να επισκευάζεται. Ιδάλλως ο καταναλωτής θα μπορεί να μεταβαίνει στη δεύτερη βαθμίδα της ιεραρχίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. And maybe if I could ask the Commission to send to members. Ναι, θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να στείλει στα κράτη-μέλη κάποια links για το πώς θα μπορούν για να, για να μπορούν να δημοσιοποιήσουν εν την έρευνα γιατί τα, κράτη, τα, μέλη μπορούν να δημοσιοποιήσουν την έρευνα μόνο όμως αν τους τα σχετικά links αν δεν έχουν τα links δεν είναι τόσο εύκολο να διαδώσουν την πληροφορία αυτή. Όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε και να διαδίδουμε πληροφορίες εφόσον τις λάβουμε Ευχαριστώ. Το επόμενο ζήτημα είναι η έκθεση από τη Λάρα Κόμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση Άμυνας. Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση είναι το σχέδιο γνωμοδότησης. Ο κ. Χέρντ από την Άλντε είναι ο εισηγητής. Ο κ. Πάιτ κυρίας Κόμη. Η κυρία Κόμη έπρεπε να συντάξει την γνωμοδότησή της ως τις 6 Ιουλίου. Υπάρχουν και γνωμοδοτήσεις από την Επιτροπή Δημοσιονομική αλλά και την ΔΕΦΚΟ. Η κυρία Κόμη λοιπόν να ανοίξει τη συζήτηση για την γνωμοδότησή της παρακαλώ. Η Λάουρα Κόμη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι Πολλέ επιτροπές ασχολούνται με αυτό το ευαίσθητο ζήτημα. Παρά τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα, η πολιτική, ασφα... πολιτική ασφάλειας και άμυνα δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Ε, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικέ βελτιώσεις. Θεωρούμε ότι το θέμα αυτό είναι υψηλή ευαισθησία μετά από τι τρομοκρατικέ επιθέσει ε, που έλαβαν χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ως Επιτροπή λοιπόν Εσωτερικής ε, Αγοράς θεωρώ ότι είναι απολύτω απαραίτητο να προτείνουμε μια σειρά ερωτημάτων που αφορούν ε, τόσο τη βιομηχανία εντός της αγοράς μας αλλά και μια σειρά δραστηριοτήτων ε, για μέγιστο διαμερισμό των πληροφοριών. Πράγματι θα υπογράμμιζα τα εξή σημεία, τα οποία θα συμπεριλάβουμε σε μια πρόταση που θα στείλουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Πρώτα απ' όλα να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της ε, κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, να δώσουμε δηλαδή στους πολίτες όχι μόνο την εντύπωση, αλλά μια πραγματική ασφάλεια και πραγματική ε, πρόληψη, να ενισχύσουμε τις αμυντικές δυνατότητες ε, μέσω της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ε, στον τομέα αυτό. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να προχωρήσουν η έρευνα και η ανάπτυξη στον τομέα προς όφελος της πρόληψης αλλά και της ανάπτυξης αμυντικών όπλων ή εργαλείων. Να θυμίσω ότι εμείς σε όλες τις περιπτώσεις είμαστε υπέρ της ειρήνης. Όπως είπα προηγουμένως, ε, διάφορες χρηματοδοτήσεις, ε, έβρεξε χρήματα θα έλεγα, ε, σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς θέλουμε ένα έργο μακροχρόνιο με υποστήριξη από τον προπολογισμό, σε μια ειδική γραμμή του προπολογισμού, πρέπει να διαρθώσουμε και να δομήσουμε μια μόνιμη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, όπου συχνά δεν υπάρχει διάλογο ούτε ανταλλαγή πληροφοριών, ειδικότερα όσον αφορά άτομα ή οργανισμού που παρουσιάζουν πρόβλημα ή που έχουν τρομοκρατικέ δραστηριότητε και μπορεί να αποτελούν σημαντική απειλή προ εμά. Όλε αυτέ οι απειλέ σχετίζονται βεβαίως με το Ισλαμικό κράτος, αλλά και με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Ε, γιατί πέραν της εσωτερικής αγοράς έχουμε και τα εσωτερικά σύνορα επίσης, ε. να καταπολεμήσουμε την παράτυπη μετανάστευση μέσω, του ελεγχού, μέσω της βοήθειας πληροφορικής. Ε, κάτι άλλο πολύ σημαντικό που ακούγεται πολύ και από την Κομισιόν και από τα κράτη-μέλη είναι ο κοινό Ευρωπαϊκός Στρατός. Αναφέρθηκε πέρυσι, ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Γιούνκερ, αλλά απαιτεί και κοινέ μυστικές υπηρεσίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταργήσουμε τις μυστικές υπηρεσίες των κρατών καθόλου. Σημαίνει ότι θα πρέπει να βρούμε ένα σημείο συνεργασίας σε συγκεκριμένα θέματα όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η τρομοκρατία. Δηλαδή να περιορίζεται αυτή η μυστική υπηρεσία σε αυτούς τους δύο τομείς. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει συστήματα πληροφορικής ε, ε, καινοτόμα υψηλής τεχνολογίας. Αλλιώς καταλήγουμε να χρησιμοποιούμε όλοι διαφορετικά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί διαφορετικά και δεν μας βοηθούν στην πρόληψη ούτε στην προστασία και στην αντίδραση σε πιθανές μελλοντικές επιθέσεις. Εγώ έχω απολύτη συνείδηση του γεγονότος ότι αυτή η στόχη είναι φιλόδοξη. Ωστόσο είμαι πεπισμένη ότι είναι εφικτή, υλοποιήσιμη στόχη, τους οποίους πρέπει να επιτύχουμε στο άμεσο μέλλον. Δεν θέλω εθνικοί εγωισμοί κρατών μελών που κάθε φορά ε, μπλοκάρουν πολλές από τις οδηγίες και τους κανονισμούς μας ε, να μπορέσει να υπερισχύσουν σε αυτή την Επιτροπή είμαστε η πραγματική καρδιά της Ευρώπης αλλά πρέπει να το αποδείξουμε με έμπρακτα και πρέπει επιτέλους για μια φορά οι εθνικοί εγωισμοί δεδομένων όλων των νεκρών που είδαμε και όλων των βομβιστικών επιθέσεων που έπληξαν ορισμένα κράτη-μέλη να μπουν λίγο στο πλάι και να καταλήξουμε να σκεφτόμαστε όλοι με ευρωπαϊκό πνεύμα. The socialist shadow is Maria Grappini, is that correct? Or is anybody else? Σκιώδης είναι η κυρία Γραπίνη, σωστά, ή θα μιλήσει κάποιος άλλος από τους σοσιαλιστές. Όχι. Έμα Μακλάρκιν, από το uh, ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την εισηγητρία για την γνωμοδότησή της. Θα ε, προσπαθήσω να είμαι όσο πιο άμεση γίνεται όσον αφορά τα σχόλιά μου όταν ε, πρωτοδιάβασα τη συγκεκριμένη ε, αναφορά στην ΙΜΚΟ ε, μου άρεσε πολύ διότι φοβήθηκα ότι θα ασχολούμασταν κυρίως με τις προμήθειες το οποίο αφορά την ΙΜΚΟ ίσως να βελτιώνουμε τον ανταγωνισμό στην ε, βιομηχανία άμυνας. Όμως αναφερθήκατε και στο ζήτημα της ε, διαφάνειας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στη συγκεκριμένη βιομηχανία και ίσως να βελτιώσουμε ε, και, την, και τις δυνατότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αμυντικού τομέα και να βελτιώσουμε την κατάσταση στον τομέα άμυνας, ενώ έχουμε θέσει και στρατηγικές για ε, την ε, οδηγία όσον αφορά τις, ε, τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Όμως όλα αυτά καλύπτονται διότι αφού αναγνωρίσαμε τη σημασία της εσωτερικής αγοράς η συγκεκριμένη γνωμοδότηση δεν συγκρατήθηκε και τελικά κάλεσε για έναν ευρωπαϊκό στρατό. Έτσι είναι η κατάσταση. Μπροστά μας ένας ευρωπαϊκός στρατός είναι μια τρομερή εισβολή στην ανεξαρτησία των κρατών ε, μελών και κατά τη γνώμη μου να δίνεται μια τέτοια άποψη από την πλευρά της ΣΥΜΚΟ είναι υπερβολικό ε, και ε, ξεπερνά το εύρος της συγκεκριμένης επιτροπής επεμβαίνοντας σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας και άμυνας η συγκεκριμένη Βουλή λοιπόν δεν έχει την εντολή να, κάνει μια τέτοια, να δώσει μια τέτοια εντολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, επίσης δεν έχει την εξουσία ε, να ασχοληθεί με ζητήματα ε, άμυνας και στρατού παρά μόνο άμα το ζητήσει το Συμβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι χάνουμε μια σημαντική ευκαιρία να επικεντρωθούμε πραγματικά σε το μίσο που έχουμε τη δικαιοδοσία και μπορούμε να βελτιώσουμε την αγορά. Καλωσορίζω λοιπόν ε, την μια υιοθέτηση των αρχών που παρουσιάστηκαν όπου ε, θα ασχοληθούμε με ζητήματα της ασφάλειας, της παροχής, ε, το μίσο που γενικά η εσωτερική αγορά, η Επιτροπή μας μπορεί να κάνει περισσότερα υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για συμβόλαια, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και θα πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ε, και να ενθαρρύνουμε τέτοιες δράσεις ε, για την έρευνα στην άμυνα και ευελπιστώ να κάνουμε, ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα για, τα, για τη βιομηχανία την οποία χρειαζόμαστε άμεσα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για το ECR αλλά και για εμένα να αποφύγουμε την αναγνώριση και την επανάληψη άλλων διεθνών προσπαθειών ιδιαιτέρως αυτών ε, που προέρχονται από το ΝΑΤΟ. Η στρατηγική αυτή λοιπόν δεν θα πρέπει ε, να ασχολείται με τέτοια ζητήματα και να επαναλαμβάνει ε, αλλά και ε, να επαναλαμβάνει ζητήματα τα οποία αφορούν την ευρωπαϊκή άμυνα. Θα πρέπει επίσης να τηρηθούν οι οικονομικές δεσμεύσεις όταν έχουμε τόσα σημαντικά ε, προγράμματα τα οποία γίνονται ταυτόχρονα. Καλό λοιπόν να υπάρξουν αλλαγές σε αυτή τη γνωμοδότηση και να επικεντρωθούμε στην αγορά για να ενισχύσουμε και να αναπτύξουμε τη βιομηχανία και τον τομέα άμυνας και ευελπιστώ ότι θα επικεντρωθούμε στο να συμπεριληφθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και ότι θα ε, περιοριζόμαστε στη δικαιοδοσία μας. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να επαναεπικεντρωθούμε πάνω σε αυτή τη γνωμοδότηση και να ε, έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα λάβει την υποστήριξη όλων μας. Um, Ευχαριστώ ο Μάρτιν Λόκερ Κύριος Ναι, θα μιλήσω εγώ στο όνομα του Μόρτιν Λόκεργαρντ. Είναι πολλές οι απόψεις ε, και ποικίλουν, αλλά γενικά είναι σημαντικό να διατηρήσουμε κατά νου τις ε, μας ε, στα πλαίσια της ΣΥΜΚΟ, δηλαδή στο θέμα των προμηθειών. Έχουμε κάποιες προτάσεις να κάνουμε για την ενίσχυση της διατύπωσης. Λαμβάνοντας υπόψη το, το δανέζικο opt-out και βεβαίως ε, σεβόμενοι ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από κόμμα σε κόμμα, θεωρεί ο συνάδελφος ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ζητήσουμε τη δημιουργία, ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, συγγνώμη, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να ζητήσουμε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού στρατού. Θέλει να διαγραφεί λοιπόν αυτό το σκέλος του κειμένου ή, εν πάση περιπτώσει, να νερωθεί κάπω η εν να νερωθει καπω η διατυπωση Μάλιστα. Εύελιν, θες να μιλήσει το όνομα της Μαρία Καπίνη. Ευχαριστώ. Η ε, συνάδελφο κυρία Γραπίνη δυστυχώ δεν μπορεί να είναι εδώ, γι' αυτό το λόγο μου έδωσε ένα σημείωμα το οποίο θα σα διαβάσω στα αγγλικά. Διότι μου είναι δύσκολο και πολύπλοκο να μεταφράζω ταυτόχρονα στα γερμανικά. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τη Λαρακόμη για το σχέδιο κειμένου και τις ε, τροπολογίες. Ε, Εμεί θέλουμε να, ε, θέλω να, συμπερι, να συμπλάβω τι εξή πτυχέ. Η Μαρία θεωρεί ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κατακαιρματισμό, ε, ο επίμονο κατακαιρματισμό τη αγορά και ότι πολλά από τα συμβόλαια συνάπτονται σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ίση πρόσβαση σε όλε τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει στην αγορά αυτή. Οι μικροπιστέ επιχειρήσει πρέπει να αντιμετωπίσουν πρέπει να ξεπεράσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για την πρόσβαση στην αγορά, ιδιαίτερα για τις αμυντικές ε, προμήθειες, είναι σημαντικό λοιπόν να, να υπάρχουν ποιοτικές και σαφείς πληροφορίες που δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις ε, στους διάφορους τομείς να εκλεπτούν τις ευκαιρίες και να παίρνουν ενημερωμένες αποφάσεις. Χρήσιμο θα ήταν να ζητηθεί από την Κομισιόν να αξιολογήσει κατά πόσο οι στόχοι της οδηγίας και του συντονισμό των διαδικασιών σε ό,τι αφορά την, ε, ε, τις συμβάσεις αυτές ε, των αμερικών προμηθειών έχουν ληφθεί υπόψη και να εξεταστεί κατά πόσο πρέπει να επικαιροποιηθεί η νομοθεσία ανάλογα με τι ανάγκε τη αγορά άμυνα. Επίση, πρέπει να εθαρρύνουμε την Κομισιόν να δώσει μεγάλη έμφαση στην έρευνα ε, και να χρηματοδοτήσει για να μπορέσουν να προχωρήσουν να προχωρήσει και η έρευνα ε, τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα της έρευνας πρέπει να θεσπιστούν όπου αυτό είναι εφικτό για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η πρόσβαση ε, να είναι πιο εύκολη στις διάφορες διαγωνισμούς για δημόσιες προμήθειες και να εξασφαλίσουμε επίσης υψηλά στάνταρτ. Επίσης πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει ανάγκη μιας, ε, ενός εξχρονισμού μάλλον του εξοπλισμού από τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα στα πλαίσια των μεγάλων δημοσιονομικών περικοπών σε μια σειρά από τομείς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η CSDP δίνει μεγαλύτερη ευελιξία, το, το πλαίσιο για τη μόνιμη συνεργασία πρέπει να είναι ανοιχτό σε όλα τα κράτη-μέλη. Ένα, δεν γίνεται αναφορά στο κοινό και κέντρο έρευνας. Ζητεί λοιπόν η συνάδελφος να γίνει μια διευκρίνηση προς την κατεύθυνση αυτή. Οι προτάσεις σε ό,τι αφορά ε, την, ε, ευρωπαϊκή, τον ευρωπαϊκό στρατό, την ενίσχυση του κλάδου ε, της άμυνας και της σχετικής βιομηχανίας, εδώ πρέπει να δώσουμε δυνατότητα σε όλα τα κρατη να βελτιώσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες. Συγγνώμη αν δεν τα είπα όλα όπως έπρεπε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Τζούλια, για τους πρασίνους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, εκ μέρου του κ. Σόλτε, του Σκιώδου, ο οποίο ζητά συγγνώμη γιατί έπρεπε να είναι παρόν σε μια άλλη επιτροπή. Γενικά, η γνωμοδότηση τη κυρία Κόμη για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση κινείται προ την κατεύθυνση που υποστηρίζουν οι πράσινοι. Στο παρόν σημείο, θέλει ο κ. Σόλτε να επισημάνει κάποια πράγματα. Οι πράσινοι συμφωνούν με τη θέση τη εισηγήτρια ότι χρειάζεται πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, ο κ. Σόλτη θα ήθελε να προσθέσει ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνεια όσον αφορά τι σχέσει μεταξύ των εθνικών αμυντικών διοικήσεων και τη αμυντική βιομηχανία. Μέχρι που θα τολμούσε να πει ότι υπάρχουν και περιπτώσεις διαφθοράς με υπερβολικό κόστος για τους φορολογουμένους. Συνεπώ η διαφάνεια είναι ύψη στη σημασία ώστε οι δαπάνε να βρίσκονται υπό τον κατάλληλο έλεγχο και να μην ε, αποφεύγονται υπερβολικέ και περιττέ δαπάνε. Επίση ο κ. Σόλτε υποστηρίζει στο τέταρτο σημείο τη νομοδότηση την εισηγήτρια όπου αναφέρεται η συμπουδαιότητα των προμηθειών. Ο μηχανισμό προμηθειών θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συνεργασία, θα βοηθήσει την καταπόλεμηση τη διαφθορά και θα βοηθήσει στη λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Ε, στο πλαίσιο της Αμυντικής Ένωσης. Θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες για ενίσχυση ε, αυτής της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ. Η κυρία Τροσέσκη, θέλετε να μιλήσετε? Όχι. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να μιλήσει για το ζήτημα αυτό? Ωραία, ξαναπαίρνω εγώ το λόγο μια έκκληση ξανά. Σας παρακαλώ προσπαθήστε ας προσπαθήσουμε να παραμένουμε εντός των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές τσακώνομαι πολύ έντονα για ζητήματα αρμοδιοτήτων μας και όταν συμβαίνει αυτό άλλοι πρόεδροι άλλων επιτροπών με κατηγορούν ότι πολλές φορές όταν εμείς γράφουμε εκθέσεις ε, πηγαίνουμε, επεκτείνομαστε σε άλλους τομείς που δεν είναι της αρμοδιότητάς μας και έτσι είναι πολύ δύσκολο για μένα να υπερασπιστώ το ρόλο της ΣΥΜΚΟ για ζητήματα που είναι της αρμοδιότητάς μας. Ξέρω ότι είναι πολλά τα ευαίσθητα ζητήματα, πολλές ε, και διαφορετικές οι απόψεις. Δεν θα τα αναφέρω λεπτομερώς, αλλά σας παρακαλώ Λάρα, ξέρω ότι θέλετε να κάνετε κάποιες πολιτικές δηλώσεις για το θέμα αυτό, αλλά δυσκολεύεται το έργο μου ως Πρόεδρο της Επιτροπής ε, αν πρέπει κάθε φορά να βρίσκουμε σημεία όπου έχουμε επεκταθεί πέραν των αρμοδιοτήτων μας. Ειδικότερα όταν γνωρίζω ότι πρόκειται πιθανότατα να κάνουμε ένα μεγάλο τσακωμό με την Επιτροπή ΣΕΝΤΕ για το ζήτημα των προμηθείων στον ε, τομέα της άμυνας. Επειδή τα αρχαία αυτά ε, ε, είχε στα χέρια τη ΣΥΜΚΟ και πρέπει να παραμείνουν στα χέρια τη ΣΥΜΚΟ. Οπότε πρέπει να φροντίσουμε να μην ξεχνάμε να εστιαζόμαστε στα ζητήματα τα οποία είναι αποκλειστικά τη δική μα αρμοδιότητα. Κύριε Ακόμη, ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θεωρώ ότι η Επιτροπή Εσωτερική Αγορά μερικέ φορέ ε, δεν έχει ξεκάθαρε αρμοδιότητε. Είναι δύσκολο να οριστούν και φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι και για σας διότι όταν μιλάμε για την εσωτερική αγορά, την κυκλοφορία των ανθόμων, των αγαθών και την κυκλοφορία και των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών, είναι δύσκολο να καταλάβουμε τι είναι αρμοδιότητά μας και τι δεν είναι, πέραν όλων των υπηρεσιών και όλων των υπολείπων πραγμάτων. Εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι μια πολύ δική περίπτωση. Δεν μιλάμε για την οδηγία για τις υπηρεσίες, ούτε για τη μια άλλη οδηγία όπου μπορεί, οποιαδήποτε οδηγία όπου μπορεί να γίνει μεγάλη συζήτηση για τις αρμοδιότητες. Εδώ μιλάμε για ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι εσωτερική. Είναι αφορά εν γενός την επικρατειά μας. Δεν είναι λοιπόν ότι εδώ υπερβαίνουμε των αρμοδιοτήτων μας, υπερβαίνουμε τις αρμοδιότητές μας. Καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση ότι γίνεται μια συζήτηση λίγο σουρεαλιστική κιόλα ε, ενώ είδαμε να υπάρχει το Brexit και ταυτόχρονα έχουμε βουλευτές που συζητούν αυτή τη στιγμή ε, θέματα τα οποία δεν θα εφαρμοστούν σε αυτούς. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να εξετάζουμε και σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Κατά τα άλλα είμαι απόλυτα στη διάθεσή σας για να αναλύσουμε το ζήτημα των ε, διαγωνισμών για τις δημόσιες προμήθειες, να εξετάσουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν την εσωτερική αγορά, αλλά το θέμα του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών, λυπάμαι, αλλά εντάσσεται στις αρμοδιότητές μας γιατί μιλάμε για ε, ε, συνεργασία αμυντική, στρατιωτική και μυστικών υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών και όχι εκτός αυτών. The deadline for amendments is the 7th of September. 7 Σεπτεμβρίου είναι η διορία Τετάρτη ε, για την κατάθεση τροπολογιών και τότε όλοι θα μπορέσουμε να σκεφτούμε και να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα ακολουθήσει μια ψηφοφορία στις 11 Οκτωβρίου. Το επόμενο κομμάτι της ημερήσιας διάταξης αφορά την ψηφοφορία στις 4 και 4. Θα περιμένω μέχρι τις 4 και μισή, ε, μέχρι ότου να έρθουν όλα τα μέλη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, το πρώτο ζήτημα με το οποίο θα ψηφίσουμε είναι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το έτος 2017. Ο Γιάκο Ψάρη είναι ο εισηγητής. Θα πρέπει να ψηφίσουμε ε, με βάση το κατάλογο ψηφοφορίας όλες οι αυξήσεις τους από μία θα διαβάσω τώρα 6612 είναι ο πρώτος αριθμός και μετά θα ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές. Λοιπόν, 6612. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6613 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6614 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6615 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 6 0 0 πρώτα τα ψηφίζουμε επί των σχολείων υπέρ κατά αποχές τα σχόλια απορρίπτονται καταπίπτουν Υπέρ ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6601 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6603 επί των σχολείων πρώτα ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται καταπίπτουν τώρα επί του ίδιου του αριθμού υπέρ κατά αποχές Λοιπόν, ναι, για το 6603, επί των αριθμητικών στοιχείων ψηφίζουμε τώρα, έτσι, υπέρ. Α, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονική ψηφοφορία, μάλιστα. Επί των αριθμητικών στοιχείων, παρακαλώ. Μάλιστα, α, καταπίπτουν. 6616, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6604, τα σχόλια πρώτα για το πιλωτικό πρόγραμμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τα σχόλια και επί των αριθμητικών στοιχείων 6604 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 6602 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 6606 τα σχόλια πρώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τα αριθμητικά στοιχεία υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 6.08 επί των σχολείων υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 6.608 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6.607 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Να δούμε τώρα από κοινού ένα 8, 1, 9, 20 και 21. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 6606 επί των σχολείων, α, συγγνώμη, 6607 επί των σχολείων, υπέρ, κατά, αποχές, καταπίπτουν. 6607 επί των αριθμητικών στοιχείων, υπέρ, κατά, αποχές, καταπίπτουν. Και τώρα θα δούμε από κοινού 22, 23, 24, 25, 26, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 6605 τα σχόλια υπέρ κατά αποχές καταπίπτουν και επί των αριθμητικών στοιχείων υπέρ κατά αποχές καταπίπτουν. 6610 επί των σχολείων υπέρ κατά αποχές καταπίπτουν και επί των αριθμητικών στοιχείων υπέρ κατά αποχές καταπίπτουν. 27 και 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 09 έχει αποσυρθεί το 09. Τα σχόλιο, το σχόλιο έχει αποσυρθεί. Τώρα επί των αριθμητικών στοιχείων, επί των ποσών όπως περιπτώσει, 6609 ψηφίζουμε επί των ποσών υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται.

Συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. 9 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. Συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Καταπίπτει. Συμβασμός 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το 17 αποσύρεται. Τροπολογία ε, συμβασμός 5 εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 6 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος έχει αποσυρθεί. Τρίτο μέρος υπέρ κατά αποχές καταπίπτει νομίζω να το επαληθεύσουμε όμως. Ναι, όντως καταπίπτει. 24 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. Τελική ψηφοφορία. Μένει μια ψήφος πέρας ψηφοφορίας. Α, έχουμε άλλη μια ψήφο υπέρ. Μάλιστα. Εντάξει. Ας α, ε, περάσουμε 22, 6 και 3 για τα πρακτικά και να πούμε ότι ε, τις, δεν ε, δούλευε τη συναδέλφου το μηχάνημα για να μπορέσει να πληρώσει, να ψηφίσει, συγγνώμη. Θέλετε να αλλάξετε συσκευή, Εύα. Ίσως για την επόμενη ισοφορία να έχει σημασία. Λοιπόν, συγχαρητήρια Λίζα. Είναι δύσκολη η δουλειά αυτή για τον προπολογισμό και τι μεσονομικέ γραμμέ. Το έχω κάνει εγώ στο, και εγώ στο παρελθόν. Λοιπόν, τώρα ενιαία ψηφοφορία για τι διαθεσμικέ ε, διαπραγματεύσει σχετικά με τον έλεγχο ε, και την αγορά όπλων. Είστε στο λόγο όμως ο συνάδη, η συνάδελφος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν προχωρήσουμε στη ψήφο, θέλω να επαναλάβω τις ανησυχίες που έχω αναφέρει ήδη όσον αφορά τις επερχόμενες ε, διαθεσμικές ε, διαπραγματεύσεις. Διάφοροι μου στέλνουν ανησυχά για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η πρόταση δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Για να καθυσχαστούν αυτές οι ανησυχίες πρέπει να φροντίσουμε οι συζητήσεις μας να βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία και σωστά στοιχεία και σωστές πληροφορίες. Οπότε θέλω να παρατηρήσω την Κομισιόν να μας στείλει όσο το δυνατόν πιο ακριβείς πληροφορίες από όλα τα κράτη-μέλη όσο το το δυνατόν συντομότερο πριν αρχίσει οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση των πυροβολών όπλων ξεκινώντας έτσι διαπραγματεύσεις που δεν θα τιμωρήσουν τελικά τίμιους πολίτες. Ευχαριστώ. Um, uh, Σημειώνω ότι ο κ. Αλά από την Κομισιόν βρίσκεται εδώ και το σημείωσε, σημείωσε τα σχόλιά σα. έχουν συμπεριληφθεί και στα πρακτικά. Κυρία Κέπαρτ, παρακαλώ. Ε, θα μπορούσα επίση εκ μέρου του κυρίου Κονφεράτη να θέσω ένα ακόμα ερώτημα ε, προ την Κομισιόν ε, για να μπορέσει να μα δώσει μια καλή απάντηση όταν θα μα απαντήσει γραπτό. Στα αγγλικά λοιπόν είπε ποιε κατηγορίε χρηστών χρησιμοποιούν αυτέ τι κατηγορίε πυροβόλων όπλων και για ποιες γνωρίζετε. Εφόσον λοιπόν έχουμε μία σειρά εξεράσεων, το συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να είναι σημαντικό για να καταλάβουμε ποιοι χρήστες θα επηρεαστούν από τα νέα μέτρα τα οποία έχουμε προτείνει. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό για το γεγονός ότι δεχόμαστε έντονη πίεση και lobbying από διάφορους ανθρώπους διότι ε, στο ίντερνετ κυκλοφορούν λανθασμένες φήμες, γι' αυτό το λόγο καλό θα είναι να έχουμε εμείς τις σωστές απαντήσεις. Να υπενθυμίσω στην Κομισιόν, στο κοινό και στα μέλη ότι πριν από την ψηφοφορία στην ΕΜΚΟ έγραψα στην Κομισιόν εκ μέρους των σχεδόν εισηγητών ζητώντας συγκεκριμένες πληροφορίες για τα θέματα αυτά καθώς και στοιχεία. Πραγματικά δεν έχουμε λάβει τίποτα. Ούτε συγκεκριμένες πληροφορίε για συγκεκριμένους τύπους ε, πυροβολών που θα συμπεριλαμβάνονται, ούτε νούμερα. Ξέρουμε ότι εσείς έχετε επαφές στα κράτη-μέλη, αναμένουμε να μας έρθουν αυτές οι πληροφορίες, θα το παρακολουθούμε και δεν θέλουμε μόνο νούμερα, θέλουμε πολύ συγκεκριμένες ειδικές πληροφορίες. Το έχουμε καταστήσει σαφές ότι είναι ζωτική σημασία ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε στο πλαίσιο οποιοδήποτε τριμερούς διαλόγου τα ζητήματα αυτά. Και βλέπω να μου γνέφουν πολλά μέλη εδώ στην αίθουσα. Αυτά λοιπόν να καταγραφεί στα πρακτικά και η Κομισιόν να είναι ενήμερη ότι ακόμα δεν μας έχει στείλει τις λεπτομερείς πληροφορίες. Έχοντας όλα αυτά υπόψη, ας ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ξεκινάμε την ψηφοφορία για τις διαθεσμικές διαπραγματεύσεις στην ομάδα και την εντολή της. Έχουμε ακόμα μια ψήφο εδώ. Ωραία, ευχαριστούμε εγκρίνεται με 24 ψήφους, 3 ε, κατά και 5 αποχές. Ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω τους παρόντες αν κάποιος από τους κοιόδης θέλει να συναντηθεί μαζί μου την επόμενη εβδομάδα παρακαλώ γνωρίστε το μου. Ladies can I ask you, is it quite cold in the... Κυρίες και κύριοι, να σας ρωτήσω, κάνει κρύο. Ναι, εδώ μες στην αίθουσα. Άκουσα παράπονα για τη θερμοκρασία της αίθουσας. Μπορείτε να το πείτε στο προσωπικό συντήρησης. Δεν είναι ότι απλά ήρθαμε από θερμά κλίματα και από τις διακοπές. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον κλιματισμό. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη αφορά το Ευρωπαϊκό Εξόμενο για το Συντονισμό της Οικονομικής Πολιτικής ε, με συντάτρια της γνωμοδότησης την κυρία Στάιλερ. Όμως ε, δεν είναι η Λούση Άντερσον η γνωμοδότρια. Υπήρξε μια αντικατάσταση. Η Καθρίν αντικαθίσταται από τη Λούση. Έχουμε 52 διαφορετικές ε, τροπολογίες και θα δώσω το λόγο κατευθείαν στη Λούση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, δεν είμαι η γνωμοδότρια, αντικαθιστώ την Κάθριν, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να, να βρίσκεται ανάμεσά μας, όμως χαίρομαι που μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της, ε, αλλά και των σοσιαλιστών. Η γνωμοδότηση, όπως γνωρίζετε, αφορά μια ε, συνεισφορά ε, σχετικά με τις ε, προτεραιότητες για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η Κάθριν θα ήθελε να πει κάποια πράγματα σχετικά με τις τροπολογίες. Θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους σκιώδεις για την συνεισφορά τους Υπήρξαν συνολικά 62 ε, τροπολογίες όπου αναφέρθηκαν ε, τα ζητήματα τα οποία ε, συμπεριλήφθηκαν στην γνωμοδότηση καθώς επίσης και επιπρόσθετα. Τα βασικότερα ζητήματα αφορούν την φορολόγηση η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει το ζήτημα της, του ΦΠΑ την ανάγκη να επιταχύνουμε την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φόροαποφυγής και επαναλάμβαμε την ανάγκη να υπάρξει εφαρμογή της νομοθεσίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για για το εξάμεινο, καθώς επίσης και να ξεκινούν διαδικασίες που παραβάσει όπου είναι αυτό αναγκαίο. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση αλλά και διαβίου εκπαίδευση, ε, πρακτικές ε, και, τέτοια, και παρόμοιες ευκαιρίες η εισηγήτρια προσπάθησε να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερε γνωμοδοτήσει ε, σε συμβιβαστικέ Οι πρώτε αποστάλησαν στου Σκιώδης σήμερα το πρωί και η Κάθριν ελπίζει ότι αυτό θα μα δώσει χρόνο στου Σκιώδης ούτω ώστε να σκεφτούν συμβιβαστικέ και ε, αδειμονεί να υπάρξει διάλογος πάνω σε αυτό στις επόμενες συνδύσεις των σκιώδων που προβλέπονται αυτήν την ε, Τετάρτη στην αίθουσα ASP 3.3 και πιστεύω ότι στην ακρόαση ε, της ΣΥΜΚΟ για τις 23 Σεπτεμβρίου θα μπορέσουμε να το εξετάσουμε λεπτομερέστερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει αντικατάσταση για τον Άνταμ Σίμφελτ. Δεν είναι. Ο Άνταμ Σίμφελτ δεν μπορούσε να έρθει σήμερα ήρθε σε επαφή μαζί μου όμως και μου ζήτησε να διαβάσω εγώ αυτά που έχει να πει και θέλει να πει τα εξής ο συνάδελφος. Όπως ελέγχθη κατά τη διάρκεια των προηγούμενων συζητήσεων που είχαμε, η ομάδα μας, το ΕΛΚ, συμφωνεί με τη θέση του εισηγητή για μια σειρά από σημεία που περιλαμβάνονται στο σχέδιο έκθεσης. Δηλαδή θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις τροπολογίες και τους ενδεχόμενες, τις ενδεχόμενες συμβαστικές προτάσεις που θα έρθουν να ενισχύσουν το βασικό μήνυμα ε, του, ε, της έκθεσης, δηλαδή τη σημασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τη σημασία του να υπάρχουν εξειδικευμένες συστάσεις αναχώρα. Είναι κάτι που θα βοηθήσει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η ευρεία υποστήριξη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι επίσης σημαντική καθώς και η υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, των start-up. Συχνά αυτές οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν διοικητικά εμπόδια. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε την οδηγία για τις υπηρεσίες, την αναγνώριση των δεξιοτήτων, την πρόσβαση στα κλειστά επαγγέλματα σε κάποια κράτη-μέλη και να εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά θα λειτουργήσουν ορθά. Χρειαζόμαστε μια, και μια ενιαία ψηφιακή αγορά. Υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου θα πρέπει να επικεντρωθούμε περαιτέρω. Θα υποβληθούν τροπολογίες στη συνέχεια τις οποίες θα υποστηρίξουμε. Σήμερα, εφόσον ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τύποι προστατευτισμού, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια ευρεία υποστήριξη για την ενιαία εσωτερική αγορά. Και οι συστάσεις που αναφέρονται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δείχνουν ότι σε ό,τι αφορά τα νομοθετήματα, η εφαρμογή είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα. Πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που μας δίνει η γνωμοδότηση αυτή για να υπογραμμίσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για τα κράτη-μέλη. Ο κύριος Σάινφερντ μου ζήτησε επίσης να πω ότι πρέπει βεβαίως να συνεργαστούμε όλοι για να πετύχουμε το στόχο αυτόν και θα υποβληθούν και ε, τροπολογίες συμβιβασμού. Ο κ. Σάνιφερ θέλει να ευχαριστήσει όλους για τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Ο Ντάν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Βίκη. Θα μιλήσω εκ μέρους του Ρίτσαρτ Σολίξ και όδους που δεν μπορούσαν να είναι εδώ σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την εισηγητρία για το έργο τη. Με πολλά συμφωνεί στο σχέδιο γνωμοδότηση, στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που είναι αδύναμη από το 2011 τότε είχε ποσοστό επιτυχία 40% και έκτοτε μειώνεται το ποσοστό. Πέρα των πραγματικών αναγκών και των συμφερόντων, αναλαμβάνει νέε εξουσίε η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει να επιλύσει όλα τα πιθανά προβλήματα. Εγώ με τι ότι πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο στην εσωτερική αγορά και λιγότερο στα προβλήματα που μπορούν να λύσουν οι ίδιε οι χώρε από μόνε του. Και αυτό σύμφωνα με τι αρχέ πάνω στι οποίε ε, έχει οικοδομηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και που περιλαμβάνονται στι συνθήκε. Σε περίπτωση προβλημάτων υλοποίηση των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στα κράτη-μέλη, πρέπει να γίνεται αξιολόγηση ώστε να εντοπιστούν οι λόγοι. Αν μία από αυτές τις η είναι οι ταχαίως επεκτηνόμενες ε, απαιτήσει για τα κράτη-μέλη, ε, πρέπει να εξευρεθούν τρόποι ε, βελτίωσης. εκφράζει ανησυχίες όσον αφορά τη σωστό εξυγχρονισμό της δημοσίας υπηρεσίας, καλωσορίζει την ψηφιοποίηση της δημοσίας διοίκησης, αλλά τονίζει ότι οι πρακτικές σε πολλά κράτη-μέλη δείχνουν ότι η ποιότητα και η διαφάνεια πρέπει να είναι προτεραιότητα και όχι η ταχύτητα. Θέλει επίσης να υπογραμμίσει ότι πρέπει να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος στα κράτη-μέλη Αλλιώ υπάρχει κίνδυνο η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπονομεύσει την οικονομική επιτυχία που προσπαθεί να δημιουργήσει. Ωστόσο, ούτω ή άλλω γενικά θα συνεχίσει τη συνεργασία με το εισηγητρή και του σκιώδες. Ευχαριστώ. Άντων Σπόρα. Ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια συναδέλφοι. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους Χιώδης για το εξαιρετικό τους έργο σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Είμαι ικανοποιημένος με τις τροπολογίες που έχουν ε, ε, προταθεί και η ομάδα μου θα υποστηρίξει τις περισσότερες. Για την ομάδα ALDE είναι σαφές ότι η εσωτερική αγορά έχει τεράστια αξία αποδεδειγμένα στην τελευταία 20 αιτία για τους λαούς μας, αλλά δεν έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας. Ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα συνέπειες του αγγλικού δημοψηφίσματος και πρέπει τώρα να προσελωθούμε στη δουλειά. Συμφωνώ στην προσήλωση στην ενιαία αγορά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Υπάρχει ανάγκη ανάπτυξη αναλυτικών εργαλείων, εργαλείων ανάλυσης, συγγνώμη, για να αξιολογείται η απόδοση της αγοράς και η πρόοδος των κρατών μελών ανάλογα με τους στόχους ανακράτως. Επίσης θεωρώ ότι δεν έχουμε εστιαστεί επαρκώς στην υλοποίηση Τη νομοθεσία για την ενιαία αγορά. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υλοποιήσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για αυτό το σκοπό. Η αρχή τη αμοιβαία αναγνώριση δεν ε, αποτυπώνεται επαρκώς στο σχέδιο γνωμοδότηση, πιστεύω. Έτσι λοιπόν έχω υποβάλει διάφορε τροπολογίε προ αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζω οι συνάδελφοι να υποστηρίξουν τι περισσότερε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Um... Ευχαριστώ. Ε, από τους πράσινους, όχι τώρα, υπάρχουν άλλοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Όχι. Ρούση, θα ήθελες πάλι το λόγο. Όχι, ευχαριστώ πολύ για όλα σας τα σχόλια. Η ε, Κάθριν ε, ανυπομονεί να συναντήσει όσο το δυνατόν περισσότερες ε, ομάδες της επερχόμενης συναντήσεις. Thank you. Ευχαριστώ. time Είμαστε αρκετά μπροστά, το οποίο είναι καλό. Και το επόμενο ζήτημα και τελευταίο ε, στην ημερήσια διάταξη αφορά την έκθεση ε, για την εσωτερική αγορά σχετικά με τη διασυνοριακή φορητότητα διαδικτυακών υπηρεσιών περιεχομένου έχουν υπάρξει 257 τροπολογίες, είχαν στις 13 Ιουλίου την πρώτη συνάντηση των σκιωδών. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Παρότι η νομοθετική πρόταση για τη διασυνοριακή φορητότητα είναι αρκετά σύντομη, Υποβλήθηκαν πάρα πολλέ τροπολογίε σημάδι ότι η έκθεση απασχολεί ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο. Οι περισσότερε τροπολογίε κινούνται προ την ειδική μου κατεύθυνση και αυτό διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τη σύνταξη ευραίων συμβιβαστικών προτάσεων που πιστεύω θα βρουν όλους σύμφωνους. Πρώτα απ' όλα να επαναλάβουμε την πρόθεση η μεταρρύθμιση αυτή να μην ερμηνευτεί ως ελεύθερη διασυνορική πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο γιατί αυτό θα υπονομεύσει την αρχή της εδαφικότητας πάνω στην οποία βασίζεται η σημερινή νομοθεσία για το copyright. Επίσης είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η προσωρινή παρουσία κάποιου ατόμου σε μια άλλη χώρα ε, πρέπει να έχει προσωρινό χαρακτήρα. Με τις τροπολογίες αυτές πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε ε, παρόχους που παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες ε, να χρησιμοποιούν τον ε, ε, νομικό μηχανισμό επαληθεύοντας σύμφωνα με τους κανόνες του κανονισμού την προσωρινή αυτή διαμονή. Με την επαλήθευση αυτή συμφωνούν όλοι ότι πρέπει να περιοριζόμαστε σε συγκεκριμένο ε, πεδίο οπότε να υπάρχει αναλογικότητα και να μην συλλέγονται προσωπικά στοιχεία πολύ περισσότερα από αυτά που είναι απολύτως απαραίτητα. Πολλέ ε, διαφορέ όμω διχογνωμίε έχουμε όσον αφορά τα αποδεκτά μέσα και εκεί έχω προσπαθήσει να βρω μια συμβαστική λύση που ελπίζω να βρει σύμφωνο τους Κιώδη και του λοιπού συναδελφού. μια συμβαστική λύση που θα περιλαμβάνει μια λίστα ε, εντό του κανονισμού που θα μπορεί να τροποποιηθεί με τα εξουσιοδότηση πράξη ανάλογα με τι τεχνολογικέ εξελίξει. Αποκλείεται ωστόσο η δυνατότητα να συμπεριληφθεί μια ανοιχτή ρήτρα η οποία θα επιτρέπει τη χρήση ε, μερών που δεν έχουν καθοριστεί στη συμφωνία μεταξύ των μελών. Μια τέτοια προσέγγιση θα εξέθεται τα πιο ευάλωτα ε, μέλη και θα ήταν αδιαφανής. Όσον αφορά την ημερομηνία θέση ισχύ, πρέπει να συμφιλειώσουμε το ότι θέλουμε να δώσουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα ένα καλό μέσο στους πολίτες ε, και ότι είναι αναγκαίο να έχει κάποιο χρόνο να προλάβει η βιομηχανία να προσαρμοστεί. Ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί λοιπόν αυτό το Γιούρις εντός 6 μηνών αλλά να τεθεί σε ισχύ μετά από 12 μήνες. Πολλά κοινά είναι τα σημεία μεταξύ των ε, διαφορών ομάδων και έτσι ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε μια συμβιβαστική πρόταση χωρίς πολλές δυσκολίες. Κυρία Πάνοβα. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Τζούλο, για την πολύ καλή συνάντηση με τους σκιώδεις ε, εισηγητές που είχαμε πριν το καλοκαίρι, που μας βοήθησε να εξηγήσουμε κάπως καλύτερα τις απόψεις μας, να εξηγήσουμε το σκεπτικό των τροπολογιών μας. Επίσης υπήρξε συμφωνία ευρύτερη στη συνάντηση αυτή ότι η αρχή πρόταση της Κομισιόν ήταν καλή και ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο σε κάποιες λίγες προσαρμογές. Χαίρομαι επίσης ε, ότι υπάρχει βούληση να ολοκληρώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα με αυτό το φάκελο, έτσι ώστε να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, παντού ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χαίρουν αυτών των υπηρεσιών περιεχομένου χωρίς να του επιβαρύνουμε με περαιτέρω γραφειοκρατία και ταυτόχρονα δίνοντα τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αυξήσουν τον αριθμό των υπηρεσιών. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει αυτή η νομοθεσία να περιορίσει τη δυνατότητα, των επιχειρήσεων στο να καινοτομήσουν ή να αποτρέψεις τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ε, να αναπτυχθούν περαιτέρω, να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ε, αυτές τις υπηρεσίες. Καλό ήταν επίσης ότι έχουμε μια κοινή κατανόηση ε, σε ό,τι αφορά τα μέτρα επαλήθευσης, ότι πρέπει να είναι αναλογικά δηλαδή, ότι πρέπει να πάνε πέρα από τα αναγκαία για να επιτευθούν οι στόχοι Επίσης ε, βλέπω ότι από τα σχέδια συμβασμού που έχω μοιραστεί ότι αυτό αποτυπώνεται ε, στην εννέα νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Στην πέντε συγγνώμη. Τώρα, το κατά πόσο θα επιλέξουμε ε, πράξη κατεξιοδότηση ή συνδυασμό δύο νομοθετικών μέσων είναι κάτι που θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες. Θέλω απλώς να πω ότι ζητήσαμε γνωμοδότηση από τις ε, υπηρεσίες της EPRS για τον πιο ασφαλή τρόπο επικαιροποίησης των, μέτρων επαλή, των μέσων επαλήθευσης και να εξετάσει βεβαίως τα υπέρ και τα κατά των διαφορών προσεγγίσεων. Ε, την έλαβα σήμερα την ανάλυση και θα την εξετάσω λεπτομερώς. Ε, ευχαρίστως Ευχαριστώ να τη μοιραστούμε βεβαίως και με τους άλλους συνεισηγητές και με τον εισηγητή ε, αυτά είναι τα βασικά σημεία τα οποία ήθελα να θίξω. Βεβαίως ε, υπάρχουν και άλλα ζητήματα δευτερεύοντα που θα προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Αυτό που έχει σημασία κατ' εμέ είναι να μπορέσουμε με επιτυχία να φτάσουμε σε πολιτική συμφωνία έως το τέλος του 2016 στην πρώτη ανάγνωση. Ε, αυτό που περιμένουν από εμά είναι να κινηθούμε γρήγορα και να δώσουμε, να φέρουμε αποτελέσματα για τι επιχειρήσει μα και για τους πολίτες μας. Αυτό είναι κρίσιμη σημασία ζήτημα, να δείξουμε δηλαδή συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα του έργου μας, έτσι ώστε ε, να αντιμετωπίσουμε και την, τον αυξανόμενο ευρωσκεπτικισμό και την έλλειψη εμπιστοσύνη ε, στους θεσμούς μας. Σας ευχαριστώ πολύ και αναμένω με ανεμονησία της εργασίας μας το προσεχές μέλλον. Μάλιστα, ευχαριστώ. Νίκολα Ντάντε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους κοιόδης. Οι εργασίες αυτές ε, για αυτή την πρόταση πιστεύω όπως είπε η κυρία Πάουνοβα θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε σε ταχεία συμφωνία. Πληρούνται όλες οι συνθήκες ε, για να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας και να επιτρέψουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ε, να απολαύουν αυτά τα ωφέλη που θα προκύψουν από αυτόν τον κανονισμό. Εγώ θεωρώ κατά πρώτον ότι πρέπει να επικυρώσουμε για άλλη μια φορά τη γενική γενικότερη υποστήριξη προς την πρόταση της Κομισιόν και να βρούμε ένα σωστό συμβιβασμό για τα πιο σημαντικά σημεία. Ε, υποβλήθηκαν, όπως πάνε άπαντες, ε, πολλές ε, τροπολογίες. Εγώ υπέβαλα 27 που στηρίχθηκαν από πολλούς σοσιαλιστές συναδέλφους και από τον σκιώδη συγγετή της Επιτροπής ε, Νομικών Θεμάτων που επίσημα θα εγκρίνει αυτόν τον κανονισμό πριν την Ολομέλεια. Όσον αφορά τις τροπολογίες, θα ήθελα να υπενθυμίσω πρώτα απ' όλα ότι επιχειρήσαμε να βρούμε ορισμούς που θα διευκρινίζουν καλύτερα την συνήθη κατοικία που είναι και η εννέα κλειδί αυτού του κανονισμού πάνω στην οποία βασίζεται και το πλάσμα δικαίου και που θα επιτρέψει αύριο να παρεχτεί δυνατότητα να έχει κάποιο πρόσβαση σε περιεχόμενο στο οποίο έχει πρόσβαση στη χώρα του όταν βρίσκεται και στο εξωτερικό. Οπότε αυτό το στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και η προσωρινή παρουσία. Και αυτό είναι ένας δεύτερο ορισμό για όπου υποβάλαμε πολλές τροπολογίες και είδαμε ότι ο ε, τις έλαβε υπόψη για να καταλήξει συμβιβαστικέ ε, τροπολογίε. Και τα ζητήματα τη επαλήθευση τη κατοικία είναι επίση ένα ε, σημείο κλειδί. Οι μέθοδοι αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ε, χωρί υπερβολική συλλογή προσωπικών στοιχείων, ώστε να μην περισφρέουν στο ιδιωτικό απόρριτο των Ευρωπαίων πολιτών. Προσοχή, το έχουμε πει από την αρχή, ένα πεσμία κλειδί είναι να αποφύγουμε οποιαδήποτε παρέσφρηση μέσω γεωγραφικού εντοπισμού και οποιαδήποτε παρακολούθηση των κινήσεων ενός ατόμου εντός ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα πρέπει να αποφύγουμε οτιδήποτε τέτοιο στοιχείο που παραβιάζει το ιδιωτικό απόρριτο των Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης θέλουμε να επιβεβαιώσουμε τη δυνατότητα του opt για όλους όσοι που παρέχουν ε, περιεχόμενο χωρίς πληρωμή όπως εθνική, εθνική, ε, εθνική τηλεοπτική σταθμή επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο εξωτερικό σε πολίτες τους που ταξιδεύουν. Επίσης υποστηρίξαμε την τεχνολογική ουδετερότητα ως αρχή και την προστασία των καταναλωτών μέσω λεπτομερούς ενημέρωσης των συνδρομητών, των ε, συνθήκων εφαρμογής του online περιεχομένου, των ε, ε, όρων παροχής της υπηρεσίας, ποιες είναι οι προσφορές κτλ. όταν κάποιος βρίσκεται στο εξωτερικό. Εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να φέρουμε εις πέρας όλο αυτό το σχέδιο πολύ γρήγορα. Πρόκειται για μια μεγάλη επιχείρηση ε, διαμεσολάβησης ε, που έρχεται σε αντίθεση με τις ριζοσπαστικές ιδέες ε, του κόμματος του εισηγητή των πενταστέρων. Μας έκανε εντύπωση που είδαμε κάποιον τόσο μετριοπαθή, τόσο ήρεμο και συζητήσιμο ώστε να καταφέρουμε γρήγορα να έχουμε αυτή την ευκαιρία έτσι λοιπόν, μέσα στους ε, μήνες που θα ακολουθήσουν την έγκριση της θέσης ισχύ αυτής της πρότασης, ε, ελπίζουμε ότι θα δούμε γρήγορα αποτελέσματα. Ε, Όσον αφορά το ζήτημα των κατευσιοδότηση πράξεων, που θέτει ο ε, στι συμβαστικέ τροπολογίε. Εμεί τι μελετάμε ακόμα. Εμεί είχαμε προβλέψει μια ρήτρα αναθεώρηση πρώτα απ' όλα και πρώτη αξιολόγηση μετά από τρία χρόνια από την έγκριση της, ε, του κανονισμού, αλλά εκεί θα διατυπώσουμε τις απόψει μας, τι συζητήσεις με του άλλου ε, συνεισηγητέ. Ελπίζουμε να βρεθεί ευρεία συνένεση εντός της Επιτροπής μας, ε, να ε, συμβάλλουμε σημαντικά στο έργο της Επιτροπής Δομικών Αποθέσεων και γρήγορα να προσφέρουμε στους Ευρωπαίους πολίτες τα ωφέλη που μπορεί να προσφέρει αυτός ο κανονισμός σε όλους τους. Uh, um, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, όπως επίσης και τους συζητητές και τους κοιόδες. Ευχαριστώ πολύ για ε, τη συνεργασία ε, που έχουμε το προσχέδιο που ε, συζητούμε αυτή τη στιγμή, συμφωνώ ε, με ε, τους συνοδέλφους μου, πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες που έχουν νόμιμα αγοράσει οι καταναλωτές και πρέπει να ταξιδεύουν. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει όμως ταυτόχρονα και ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο επιβεβαίωσης αρχικά σχετικά με το αν θα πρέπει να είναι ε, μια ανοιχτή ή κλειστή διαδικασία ε, υποστήριξα μια υβριδική διαδικασία που θα προσπαθεί να ε, υποστηρίξει το συνδυασμό της ανοιχτής και κλειστής λίστας όμως δεδομένων των τρομπολογιών που έχουν κατατεθεί πιστεύω ότι είμαστε πιο κοντά στην κλειστή, στην κλειστή λίστα και θα κατευθυνθούν προς εκεί οι συμβιβαστικές διότι είναι σημαντικό η ε, μεταφορητότητα να ε, παρέχει αυτό το ε, περιεχόμενο και η κλειστή λίστα είναι η μόνη εναλλακτική για να το προσφέρει. Θα πρότεινα επίσης προς όλους σας να υποστηρίξετε τις τροπολογίες που επικεντρώνονται στην ε, διατήρηση της εντοπιότητας από έγγραφα τα οποία έχουμε δει ε, πρόσφατα ε, φαίνεται ότι προωθούν την διασυνοριακή πρόσβαση και θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, ενώψη, υπό, λαμβάνοντας υπόψη το τι ε, συνέπειες θα έχει αυτό, ε, διότι θα αντικατοπτρίζει το καλό έργο που κάνουμε στην Επιτροπή μας. με απασχολεί η τροπολογία 81 της Άλντε σχετικά με τις δωρεάν υπηρεσίες και την πληρωμή υποχρεωτικής άδειας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο όσον αφορά την ε, επιβεβαίωση, όμως δεν αντιστοιχεί ε, στις ε, επαμοιβή υπηρεσίες. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρεί αυτή τη δυνατότητα και να φαίνεται στην νομοθεσία και θα πρέπει να γίνει σε αυτό το πλαίσιο και χαιρετίζω το γεγονό ότι και άλλοι το υποστηρίζουν. Ανησυχώ επίσης ε, σχετικά ε, με, όσους, ε, με τον ορισμό αυτών οι οποίοι μένουν περιστασιακά. Θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε αυτό σχετικά με ποιους είναι μόνιμους κατοίκους και ποιους παραμένουν σε μια περιοχή για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δεν θέλουμε λοιπόν να ε, δημιουργήσουμε παραθυράκια όσον αφορά τις διασυνοριακές υπηρεσίες και γι' αυτό καλώ τους συναδελφούς να μην υποστηρίξουν ε, τις τροπολογίες που θα επιτρέψουν τέτοια παραθυράκια. Υποστηρίζουμε επίσης το πλάσμα δικαίου και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στα κράτη-μέλη όταν προσφέρουν πρόσβαση δεν θα πρέπει να ε, προσθέσουμε και άλλες υποχρεώσεις στους ε, πάροχους, όμως θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σχετικά με το να βρίσκουν ποιο είναι το κράτος μέλος όπου κατοικεί ο εκάστοτε καταναλωτές. Για άλλη μια φορά λοιπόν επαναλαμβάνω τα όσα υπόθηκαν και ότι θα μπορέσουμε ε, να ολοκληρώσουμε το συγκεκριμένο κείμενο χαιρετίζω τις ε, τροπολογίες και ανυπομονώ στην επόμενη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Η Οντίτα Σαρσέβα. Ευχαριστώ. Να ευχαριστώ και εγώ, ε, λέει η κυρία Τσαράνζοβα, ε, τον εισηγητή. Πριν μιλήσω για το σύστημα επαλήθευσης, θα ήθελα να πω ότι η ομάδα μου μπορεί να υποστηρίξει τις ιδέες που περιλαμβάνονται σε πολλές από Υποστηρίζουμε την προσθήκη μιας διατύπωσης σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτών των κανόνων σε όλους τους πάροχους, ανεξάρτητα από το ποια είναι η βάση τους, να μην αποτρέψουμε την πρόσβαση στο τοπικό περιεχόμενο, τεχνολογική ουδετερότητα, να μην οδηγήσει αυτό σε αύξηση των τιμών και η συμπέριληψη μιας ρήτρας αναθεώρησης. Σε ό,τι αφορά τώρα τις λεπτομέρειες, άρθρο 1, πεδίο εφαρμογής, εδώ ελπίζω να μην ληφθεί ε, υπόψη αυτή η προσθήκη ε, του legally required, μια σειρά από διατυπώσεις που προτείνεται να προσθεθούν εδώ, νομίζω πως δεν χρειάζονται, είναι αυταπόδεικτα αυτά, ε, δεν πρόκειται παράνομο περιεχόμενο να γίνει ξαφνικά νόμιμο ούτως ή άλλως. Αυτό είναι λοιπόν το illegal ε, content δεν έχει νόημα. Ό,τι προσθέτουμε δημιουργεί μάλλον ασάφεια. Τώρα, όπως και με το άρθρο 1 εδώ στους ορισμούς, πρέπει να προσέξουμε ε, με τον ορισμό του κράτους μέλους ε, διαμονής ή του κράτους μέλους προσωρινής παρουσίας. Δεν πρέπει να διαβρύνουμε τον ορισμό αυτό παραπάνω από όσο πρέπει, από όσο χρειάζεται. Ε, και εδώ επιμένω στην τροπολογία μου στο σημείο Γ. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο ε, να επιβληθούν περαιτέρω απαιτήσει στους παρόχους ε, και στους συνδρομητές. Ό,τι αφορά το περιεχόμενο το επιγραμμικό, εμείς δεν θέλουμε να αποκλείσουμε το περιεχόμενο το επιγραμμικό μέσω τηλεόρασης. Γίνεται αυτό στο δημόσιο επίπεδο, στο επίπεδο δημόσιας τηλεόρασης με τα χρήματα του καταναλωτή. Γιατί λοιπόν να μην το κάνει αυτό και ένας ιδιώτης. Πρέπει να θεωρηθεί πληρωμή και η άδεια η τηλεοπτική. Για το άρθρο 3, συμφωνούμε με το 3α και το 3β, ε, το opt για τι ελεύθερε υπηρεσίες, εκεί δεν συμφωνούμε, πρέπει η τηλεοπτική άδεια, περιλαμβάνω, να θεωρηθεί πληρωμή. Τώρα για την επαλήθευση, αυτό είναι το σημείο κλειδί, δεν μπορούμε να δεχθούμε το συμβιβασμό στο συγκεκριμένο άρθρο, δεχόμαστε την ιδέα ενός καταλόγου, αλλά ο κατάλογο αυτός πρέπει να είναι κλειστό, πρέπει να είναι περιορισμένο. Έχουμε συμπεριλάβει επίσης στις τροπολογίες μας κάποιες κόκκινες γραμμές κλειδιά. Πρώτα απ' όλα η παρακολούθηση ενός μια διεύθυνσης IP δεν είναι απαραίτητη και πρέπει να εξαιρεθεί. Οι διευθύνσεις IP δεν είναι ε, αξιόπιστες. Υπάρχουν μια σειρά από πρόξεις, υπάρχουν VPN που επιτρέπουν να κρύψει κάποιο στην πραγματική διάμεση. Ο κύριο και η κυρία Άρνολντ από το Κάνσα στι Πολιτείε, παραδείγματο χάρη. Η χώρα του έω πρόσφατα είχε 600 εκατομμύρια διευθύνσει IP. Είχαν ε, γι' αυτό λάβει, δεχτεί επιθέσεις, ε, ε, γράμματα μίσους, έχουν έρθει να, στο σπίτι τους για να ψάξουν παιδιά τα οποία έχουν απαχθεί ή κλεμμένα αντικείμενα. Ε, λοιπόν, η φορητότητα δεν πρέπει να μας στείλει ε, στην ε, εποχή όπου ξαφνικά οι εταιρείες μουσικής ε, έκαναν μήνυση σε γιαγιάδες με βάση λάθος IP για παράνομο κατέβασμα μουσικής. Πρέπει λοιπόν να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπίας. Θα σταματήσω εδώ, γιατί δεν έχω χρόνο. Θέλω να σας καλέσω όλους να διαβάσετε την τροπολογία μας, την 208 και τέλος να πω ότι δεν πρέπει να γίνει πιο δύσκολη η φορητότητα από το να γραφτεί κάποιος να ψηφίσει ας πούμε. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, ελπίζουμε να φέρουμε συγκεκριμένα από τα αποτελέσματα για τους συμπολίτε μας. Ευχαριστώ. Τζούλια Ρέντα. Τζούλια Ρέντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους Θεόδης ε, για όλη τη δουλειά που έχουν κάνει για αυτή την πρόταση. Δυστυχώ πολλές από τις συμβιβαστικέ ε, τροπολογίες κινούνται προς την λάθο κατεύθυνση κατά την άποψή μας και σε ορισμένε περιπτώσει ε, αποτελούν οπισθοδρόμηση σε σχέση με την αρχική έκθεση του κυρίου Σιγητή. Πολλά από τα όσα έχουν προσθεθεί στο κείμενο αυτού του κανονισμού ε, προτείνεται περισσότερο να καθησυχάσουν τους ανθρώπους. Το ανέφερε και η Δίτα, αλλά να τονίσω, όταν λέμε νομικά απαιτούμενος στο άρθρο 1, αυτό μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικά νομικά προβλήματα, διότι δεν είναι σαφές τι εννοεί τον ε, έχει εγγραφεί νόμιμα ο συνδρομητής, ε, ο καταναλωτής στην υπηρεσία και φυσικά υπάρχει υπηρεσιών. Δεν παρέχουν φορητότητα σε ανθρώπους που έχουν γραφτεί παράνομα αλλά σημαίνει επίσης ότι και ο παρόχος υπηρεσιών ε, παρουσίαζε το περιεχόμενο παράνομα γιατί δεν είχε άδεια. Μιλάμε εδώ για νομοθεσία καταναλωτών, για την οδηγία ψηφιακού περιεχομένου ταυτόχρονα που περιέχει διατάξεις για το τι υποτίθεται ότι συμβαίνει, τι δικαιώματα έχει ένα καταναλωτής σε περίπτωση που ένας πάροχος υπηρεσιών του έχει παράσχει παράνομο περιεχόμενο. Αν πρόκειται λοιπόν να βάλουμε το legally acquired σε αυτή την νομοθεσία, μπορεί να καταλήξουμε να ερχόμαστε σε αντίθεση ε, να αντιφάσουμε με την άλλη νομοθεσία ε, που μελετάμε αυτή την εποχή. Ήθελα να το τονίσω γιατί πολλέ από αυτέ τι δηλώσει που βλέπουμε. Ναι, φυσικά θέλουμε ο κόσμο να ε, τηρεί την νομοθεσία, δεν χρειάζεται να το γράφουμε σε κάθε νόμο μέσα. Το ίδιο ισχύει και για το πραγματική και σταθερή κατοικία αντί για συνήθη κατοικία ή όπως βλέπουμε στην τροπολογία 3 προσθέτουμε το προσωρινά μη μόνιμα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα είναι περιτά όλα αυτά. Κάποια σημεία που θεωρούμε την εντάξει, που είναι καλά, Το ότι δεν υπάρχει τακτική επιστροφή σε ένα κράτος ε, θεωρούμε ότι είναι καλό. Η δική μας τροπολογία 164 δεν καλύπτεται από τη συμβιβαστική τροπολογία. Η 164 προτείνει να έχει κάποιο ε, παραπάνω από ένα κράτη κατοικία. Ε, δεν υπάρχει αυτό το κείμενο στη συμβιβαστική τροπολογία, οπότε θέλουμε να ψηφιστεί ξεχωριστά. Στη συμβιβαστική 4 θεωρούμε επίσης ότι είναι καλό που ο εισηγητής προτείνει να διασφαλίζουμε ότι η φορητότητα δεν θα δημιουργεί υπεραιτερό κόστος για τους καταναλωτές και ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθείτε ως δικαιολογία αύξηση του κόστου Συμφωνούμε με αυτή τη συμβαστική τροπολογία, αλλά θέλουμε η δική μας τροπολογία για το 95 να συμπεριληφθεί. Περιλαμβάνει αυτή η τροπολογία και μια έννοια που πιστεύω έχουν συμφωνήσει όλες οι ομάδες με αυτήν, ότι ο παροχός υπηρεσιών πρέπει επίσης να μπορεί να σας παρέχει πρόσβαση και στο τοπικό κατάλογο περιεχομένου, στο χώρο που βρίσκεστε. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό και θα το επιθυμητώ από όλου να συμπεριληφθεί το περιεχόμενο αυτή τη τροπολογία. Όπω είπε η Ντίτα, η συμβιβαστική 5 περιέχει μια κρίσιμη διαταξή. Θεωρούμε ότι το κείμενο του συμβιβασμού ε, είναι αντιφατικό, διότι πρώτα απ' όλα παραθέτει τη δειγματοληπτική εξέταση των ΑΕΠ ε, ως επιλογή για να καθοριστεί ε, το κράτο κατοικία και μετά λέει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται λόγω τη δυνατότητα ε, εντοπισμού των χρηστών. Αυτό έρχεται σε αντίφαση με τη Συμβαστική 14 που αναφέρεται στην αναλογικότητα των μέσων που θα χρησιμοποιούνται. Για να συμφωνήσουμε λοιπόν με αυτή τη διάταξη, πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι είναι σημαντικό η χρήση δύο μέσων επαλήθευσης από τον πάροχο υπηρεσιών πρέπει να είναι το μέγιστο και να αποτελεί εξαίρεση, να γίνεται κατεξαίρεση μόνο από τον κανόνα της χρήσης ενός. Επίσης, η επιλογή της δήλωσης ε, κράτους κατοικίας, ε, που αν θυμάμαι καλά και στη, δεν συμπεριλαμβάνεται καν στην ε, θέση του Συμβουλίου. Είμαστε υπέρ ε, του συντομότερης υλοποίησης του κανονισμού εντός εξαμήνου και θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή, επειδή πολλά άρθρα δεν αντιστοιχούν σε συμβιβαστικές τροπολογίες αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι ο εισηγητής προτείνει να διατηρηθεί η διατύπωση της Κομισιόν. Εμείς γενικά την υποστηρίζουμε. Όσον αφορά τις αιτιολογικές σκέψεις, έχω κάποιες επίσης παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα στη συμβιβαστική 7 δεν είναι σαφές ότι η σκοπή του ταξιδιού που παρατηρείται εκεί είναι παραδείγματα. Απλά φυσικά δεν μπορούμε να παραθέσουμε όλου του πιθανού λόγου για του οποίου κάποιο μπορεί να ταξιδέψει. Ε, ε, και να έχει, έχει μια καλή αιτιολογία για να χρησιμοποιήσει τη φορητότητα. Πρέπει λοιπόν να το καταστήσουμε απολύτω σαφές ότι αυτά είναι απλά παραδείγματα ή αλλιώ να τα βγάλουμε από το κείμενο. Και τέλος, όσον αφορά τη συμβαστική 12, λέει ότι οι δικαιούχοι όχι μόνο θα πρέπει να μπορούν να επαληθεύσουν την ε, κατοικία αλλά και την προσωρινή παρουσία σε ένα άλλο κράτο μέλο. Για ποιο λόγο δικαιούχο θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να λάβει αυτέ τι πληροφορίε. Δεν υπάρχει λόγο ο δικαιούχο ενό δικαιώματο να γνωρίζει από ποιο κράτο μέλο αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο αν βρίσκεται στο κράτο κατοικία του, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα είχε πρόσβαση στο περιεχόμενο του σε άλλου. Και αν βρίσκεται σε άλλο κράτο μέλο, προσωρινά, δεν υπάρχει λόγο ο κάτοχο των δικαιωμάτων να ξέρει σε ποιο κράτο μέλο βρίσκεται και έτσι να ανοίξουμε και άλλα προβλήματα προστασία δεδομένων. Τέλο, όσον αφορά το ζήτημα του κατά πόσο οι υπηρεσίε για τι οποίε έχει ε, καταβληθεί κάποιο τέλο άδεια πρέπει να συμπεριληφθούν. Έχουμε δει ότι έχει διαρρεύσει από τις επερχόμενες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, εξάγει κανείς διάφορα συμπεράσματα. Εγώ, όπως κατάλαβα την εξαίρεση των δημόσιων ραδιοτηλεπτικών υπηρεσιών, ε, ε, μου φαίνεται σαν υπόσχεση ότι αυτό θα το αντιμετωπίσουμε στην αναθεώρηση του copyright στο άμεσο μέλλον. Οπότε δεν χρειάζεται να το δούμε εδώ. Αλλά αν δούμε τώρα τον προτινόμενο κανονισμό, που θα έρθει επιτρέπει στους ραδιοτελεπτικούς σταθμούς να βασίζονται στην αρχή της χώρας προέλευσης μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Εφόσον λοιπόν η υπηρεσία η online είναι απλά βοηθητική ως προς ε, τις υπόλοιπες υπηρεσίες, οπότε πιθανότατα δεν θα επιτρέπουν στους ραδιοτηλεπτικούς σταθμούς να ε, απαγορεύουν ε, το geo Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν διότι και οι κανόνες για την χώρα καταγωγής είναι εντελώς προαιρετικοί για τους ραδιοτηλεπτικούς σταθμούς. Αν δεν τους συμπεριλάβουμε λοιπόν στη φορητότητα, δεν θα έχουν καμία απολύτως υποχρέωση να παράσχουν πρόσβαση, ακόμη και στους δικές τους συνδρομητές από τη χώρα τους, όταν θα βρίσκονται στο εξωτερικό. Φιλίπ παρακαλώ. Merci, Madame la Présidente. Euh, tout d'abord... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τον σκιώδη εισηγητή ε, για τη δουλειά τους, για αυτό το θέμα το οποίο ασχολείται και πολύ καιρό. Τέσσερα σχόλια. Πρώτον, τα κριτήρια επαλήθευσης για την χώρα διαμονής. Τροπολογίες 8 και 12 του εισηγητή που καθιστούν υποχρεωτική αυτή την επαλήθευση και η ιδέα μιας πιο κλειστής λίστας μας φαίνεται πιο καλή η κλειστή λίστα. Και κάτι ακόμα που συνδέεται, το να συνδέσουμε, το να, το δώσουμε στην Κομισιόν από πράξη κατεξουδότηση τη δυνατότητα να τροποποιήσει τα κριτήρια, δημιουργεί πρόβλημα. Διότι εφόσον αποφασίσουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες τώρα εδώ, είναι επειδή είναι σημαντικές λεπτομέρειες, να έρθει μετά μια πράξη κατεξουδότηση και να αμφισβητήσει, να διακυβεύσει αυτά που αποφασίσαμε, εμένα με δημιουργεί πρόβλημα. Τρίτον, για τον ορισμό της προσωρινής ε, παρουσίας. Εξαιρετικά σημαντικός ορισμός, διότι επιτρέπει να αγγιηθούμε μια πραγματική, ένα πραγματικό δικαίωμα για τη φορητότητα του περιεχομένου των καταναλωτών που μετακινούνται από μια χώρα στην άλλη, χωρίς βεβαίως να υπάρξει υπερβολική διεύρυνση του πεδίου ε, του κανονισμού, ε, δηλαδή να μην παρακαμφθεί η εδαφικότητα. Είναι σημαντικό λοιπόν ο ορισμός εδώ να είναι σαφής. Η τροπολογία 67 δίνει, διευκρινίζει το μεταβατικό χαρακτήρα της προσωρινής συμφωνίας καθώς και τον 172 που αναφέρεται στο προσωρινό χαρακτήρα. Και κάτι ακόμα, για τις άδειε. Έχω την εντύπωση ότι για να μην ε, παρεμποδίσουμε Άλλε συμβασιακές λύσει στα πλαίσια των εισοδηγίας για την ε, ομαδική διαχείριση, λογική διαχείριση, είναι σημαντικό να λέει ο κανονισμός ρητά ότι δεν επηρεάζει αυτό τι άδειε σε ό,τι αφορά τη φορτότητα του περιεχομένου, δεν αφορά δηλαδή τις υπηρεσίες που προ, προβλέπουν ήδη διασυνοριακή πρόσβαση. Κάποιε τροπολογίε πρέπει οπωσδήποτε να, να στηριχθούν εδώ, οι 44, 47 και 68 μεταξύ άλλων. Ευχαριστώ πολύ. Andreas. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την κυρία Παλούβα. Θεωρώ ότι όσον αφορά τις ε, συζητήσεις ε, για την συγκεκριμένη οδηγία είναι επικοδομητικές ε, μέχρι στιγμής και για αυτό το λόγο είμαι ευγνώμων απέναντι σε όλους τους συναδέλφους και τον συνάδελφο Τσόλο, όμως θα ήθελα να σημειώσω τέσσερα σημεία ε, αντίθετα με αυτό το οποίο θα ευχόμασταν στη συγκεκριμένη οδηγία δεν πρόκειται ε, για μία επέμβαση που ξεπερνά τα σύνορα αλλά για ε, την μεταφορητότητα η οποία θα κατεστεί εφικτή και θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτά τα δύο δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Δεύτερον, υποστηρίζω ότι οι δωρεάν υπηρεσίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην οδηγία σε περίπτωση που αυτό είναι επιθυμητό. Τρίτον, είναι σημαντικό να έχουμε μια πραγματιστική και ε, λογική εξέταση του τόπου κατοικίας και αυτό μπορεί να γίνει άμεσα μέσω της εφαρμογής ε, από την ε, της εφαρμογής της μεθόδου από την πλευρά των παρόχων που είναι δουλειά τους Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα γι' αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν οι πραγματιστικές δυνατότητες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια λίστα η οποία θα μπορεί να ακολουθεί και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η ε, Παύλοβα το είπε σωστά όσον αφορά ε, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Θα πρέπει να δούμε τι λειτουργεί όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο όμως ε, στο ζήτημα της ασφάλειας θα πρέπει να προσέξουμε το θέμα της, ε, του γρήγορου και γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να περιοριστούμε χρονικά και ε, σώνει και καλά μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου να τα έχουμε συμπεριλάβει όλα. Ευχαριστώ πολύ. Από προσωπική άποψη χαίρομαι ιδιαίτερος που, έχω, που βλέπω πολλούς ανθρώπους να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη ε, συζήτηση. Είναι σημαντικό ο καθένας να έχει τα δικαιώματα μαζί του όποτε ταξιδεύει. Θα πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει με άλλες οδηγίες και θα πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια πάνω σε αυτό. Όμως πρέπει να πω ότι ε, ε, θα μπορούσα να βλέπω διάφορες ε, σειρές ε, και όταν είμαι εδώ στις Βρυξέλλες. Έτσι λοιπόν για να έχουμε αυτή τη δυνατότητα θα πρέπει να το κάνουμε. Νομίζω ότι ε, ε, εδώ κλείνουμε σε περίπτωση εκτός και αν ο κ. Ζόλου θέλει να δώσει κάποια απάντηση. Είναι πολύ γρήγορα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους για όλα τα σχόλια. Πολλές από τις αμφιβολίες που ακούσαμε θα τις ε, ξεπεράσουμε στη συνεδρίασεις μας. Επαναλαμβάνω την πρόθεσή μας το να κλείσουμε ταχαίως την έκθεση αυτή ώστε να εξυπηρετήσουμε γρήγορα τους πολίτες. Όλες οι ωφέλιμες υποδείξεις ώστε να αντιμετωπίσουμε τις περιπτώσεις κατάχρησης και να καλύψουμε τις γκρίζες ζώνες, ε, να τις ξεκαθαρίσουμε που θα οδηγήσουν σε δυσκολίες κατά την εφαρμογή του κανονισμού θα είναι ευπρόσδεκτες ε, και πιστεύω ότι έτσι θα υπερβούμε όλα τα εμπόδια. Ευχαριστώ. Excellent. The next... Um, Ωραία. Την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε το θέμα αυτό θα είναι όταν θα συζητήσουμε τις συμβιβαστικές, μερικές εκ των οποίων έχουν ε, συζητηθεί ε, σήμερα, αλλά θα ξανασυζητήσουμε για αυτές τις 22 Σεπτεμβρίου, μέχρι πριν αποφασίσουμε